Η ημερήσια διάταξη, γιατί και εγώ και το προσωπικό μου δεν έχουμε καταλάβει τι περιλαμβάνει αυτή η ημερήσια διάταξη. Περιμένω να εμφανιστούν, ξέρετε, συνάδελφοι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανυπομονησία που θέλετε οπωσδήποτε να προωθήσετε έτσι ε, τις εργασίες της Επιτροπής μας. Wir sind vor der Beendigung des Ξέρετε δεν έχει περάσει και το ακαδημαϊκό τέταρτο ακόμα. Και μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση με το επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη. Όπως αναφέρεται κύριε συνάδελφε, στην ημερήσια διάταξη, είναι η έκθεση του κυρίου Κούκαν και θα παρακαλέσω τον εισηγητή να μας ε, διαφωτίσει δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Παρακαλώ κύριε Κούκαν. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ επιβεβαιώνω ότι εσείς ήσασταν στην ώρα σας και περιμένετε τους υπολείπους να έρθουν. Για να είμαστε δίκαιοι. Τώρα, για την ε, έκθεση για το μηχανισμό γειτονίας. Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω την πολιτική σημασία αυτής της έκθεσης για τη δική μας την Επιτροπή, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, διότι εμείς είμαστε αυτοί που προσέχουμε πάντα την πολιτική γειτονία. Επιπλέον δε, οι συζητήσεις για το μηχανισμό αυτό και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτης μας δίνει τη δυνατότητα ως Κοινοβούλιο να βεβαιωθούμε ότι η χρηματοοικονομική συνδρομή στις γείτονες χώρες θα αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή η δυνατότητα μας δίνεται μία φορά στα 7 χρόνια, επομένως θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε πλήρως. Όταν προετοίμαζα το σχέδιο έξεσης, ε, ήρθα σε επαφή με αρκετούς ενδιαφερομένους ε, για το έγγραφο αυτό και από χώρες εταίρους, ε, αρχές, πρέσβεις, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ήθελα να συναντηθώ με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για να λάβω και τη δική τους τη συνεισφορά. Και μάλιστα τη συνεισφορά των ανθρώπων που ενδιαφέρονται περισσότερο για το μηχανισμό αυτό. Ε, συναντήθηκα ε, σε μια άτυπη συνάντηση, αλλά πολύ επικοδομητική, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους ε, ε, του EIS και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό. Όσον αφορά τώρα το μηχανισμό γειτονία, θεωρώ ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αντανακλά τι βασικέ προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην πολιτική γειτονία και τη συνολική πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκίνησε από πέρσι. Υπάρχουν μερικά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να χαιρετήσω ιδιαίτερα στην, ε, στον μηχανισμό αυτό. Καταρχήν, η αυξημένη συνοχή μεταξύ της πολιτικής γειτονίας και του μηχανισμού γειτονίας μέσω προγραμμάτων δράσης, ε, εγγράφων προγραμματισμού και ε, της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού σε σχέση με τον τρέχοντα μηχανισμό. αναφέρεται μια συγκεκριμένη προσέγγιση για την πολιτική γειτονία με κάθε χώρα εταίρο και γίνεται μια συγκεκριμένη διαφοροποίηση που διασφαλίζει ότι κάθε χώρα θα αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα στο βαθμό που το απαιτεί η ίδια και τις επιτρέπουν και οι δυνατότητές της. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη στις χώρες οι οποίες δεσμεύονται να δημιουργήσουν δημοκρατικές κοινωνίες και να αναλάβουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, θα ε, βοηθήσουν και θα έχουμε τις αρχές ε, της αμοιβαία λογοδοσίας. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί και ο πρόεδρος Μπροκ, ότι κάποιε από τις τροπολογίες που κατατέθησαν είναι κοινέ για όλα αυτά τα μέσα χρηματοδότησης ε, και ε, είναι κοινέ και για την κοινή προσέγγιση. Δεν θα υποσέλθω λοιπόν σε λεπτομέρειες από αυτόν και να σας πω ότι αυτή η προσέγγιση να τα εξετάσουμε όλα από κοινού είναι πολύ χρήσιμη και θεωρώ ότι θα πρέπει να τη διατηρήσουμε μέχρι τέλους. Για το σχέδιο κειμένου τώρα, να σας πω ότι εγώ θα ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση στην προσέγγιση που βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες και στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίες και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει πρωτίστως να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες να ενισχύουν τη δημοκρατία, την καλή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Και επίσης θα ήθελα να γίνει μεγαλύτερη διαφεροποίηση Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να συμπεριληφθεί στο κείμενο του κανονισμού ένα σαφή μηχανισμό για αυτή τη διαφοροποίηση. Αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να είναι η αρχή που θα διέπει το στρατηγικό προγραμματισμό, τα έγγραφα τα οποία θα διατυπωθούν για διάφορα χρόνια για αρκετέ χώρε και αυτή η αρχή θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή όλων των ε, ε, πρωτοβουλειών και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσθέρεται στήριξη σε αιτήσια βάση για τις χώρες οι οποίες κάνουν ε, προσπάθειες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν και προσπαθούν να εκδημοκρατιστούν και θεωρώ ότι χρήζουν περαιτέρω υποστήριξη από πλευράς μας. θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να αναφέρονται πολύ καλύτερα στο μηχανισμό αυτό οι εταιρικέ σχέσεις με την κοινωνία, διότι είναι στο επίκεντρο της αναθεωρημένης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Θεωρώ ότι αυτές οι συμπράξεις με την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να είναι ως βασικός στόχος του μηχανισμού αυτού και προτείνω να δοθεί ιδιαίτερος ρόλος στην κοινωνία των πολιτών και να διασφαλίσουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα λάβουμε μέτρα προκειμένου να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της κοινωνίας για να διαδραματίσει το ρόλο της κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του μηχανισμού. Κάτι τελευταίο, σας είπα προηγουμένως ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκλογικεύσει το πεδίο εφαρμογής αυτού του μηχανισμού, ώστε να υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της πολιτικής γειτονίας. Και θεωρώ ότι δεν θα ήταν δόκιμο να περιλάβουμε πάρα πολλούς επιπλέον στόχους, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος από έγγραφο προγραμματισμό να είναι ένας κατάλογος επιθυμιών, γεγονός που σημαίνει ότι θα μειωθεί η σημασία του και ο μηχανισμός ε, δεν θα είναι τόσο σημαντικός. Προσβλέπω λοιπόν στα σχόλιά σας και είμαι διατεθειμένος να συναντηθώ ε, με τους συναδέλφους και τους κοιόδης ε, εισηγητές προκειμένου να συζητήσουμε, διότι υπάρχει χρόνος και να συζητήσουμε και να τροποποιήσουμε το κείμενο για να είναι ένα ουσιαστικό κείμενο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κούκαν για την ενημέρωση αυτή. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεσή σας στην Επιτροπή μας. Θα δώσουμε στο λόγο στον κύριο Λάκη Σκιώδη, εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δεν έχω και πολλά να πω. Υποστηρίζουμε την έκθεση, είναι πολύ καλά διατυπωμένη. Ε, βλέπω ε, το χέρι του ε, Υπουργού Εξωτερικών σε αυτήν την έκθεση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σημασία που δίδεται ε, στις οργανώσεις των εργαζομένων και τα συνδικάτα, καθώς επίσης και στο ρόλο του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού και η αρχή περισσότερα για περισσότερα θα πρέπει να συνοδεύεται από την αρχή λιγότερα για λιγότερα ε, για την οποία χρειαζόμαστε πολύ σαφείς μετρήσεις, ε, benchmarks. Ε, είναι επίσης πολύ σημαντικός ο ρόλος των κατεξιοδότηση πράξεων και θα ήθελα να... και έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες για να βελτιώσουμε ορισμένα σημεία της έκθεσης που ήδη υπάρχουν βέβαια. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία παρακαλώ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε ε, Κούκαν. Κύριε Σιγητά, βλέπουμε ότι συζητήσατε πολύ για τις τροπολογίες σας. Yeah. Ε, στόχος σας ήταν να μεταφραστούν οι ε, αναθεωρισμένοι πρώτα προσανατολισμοί γειτονίες μετά από τα κινήματα εκδημοκρατισμού της νότιας όχθης Μεσογείου πριν από ένα χρόνο περίπου. Και βλέπω ότι στους στόχους σας αναφέρεται ρητά τη συμπερίληψη ενός ε, θεσμικού μηχανισμού έτσι ώστε σε όλα τα επίπεδα να συμμετέχουν οι ενεχόμενοι με τη διαφορετική μορφή κοινωνία των πολιτών, των χωρών αυτών και μάλιστα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την υλοποίηση και τον έλεγχο για την παρακολούθηση. μου επιτρέπετε θα προσπαθήσω και εγώ να εμπλουτίσω την πρόταση. Πώς θα ενσαρκωθεί να προτείνω αυτός ο μηχανισμός και να επιμείνω στη δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι χώρες αυτές ε, για την εγχώρια λογοδοσία, δηλαδή να έχουν την ικανότητα οι κοινωνίες οι ίδιες να αξιολογούν ε, τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών γειτονίας που εφαρμόζονται. Επίσης πιστεύω η αναφορά που γίνεται στη βαθιά δημοκρατία, deep democracy, είναι πάρα πολύ εύστοχη, αλλά μπορεί και ε, περαιτέρω να ενισχυθεί στις προτάσεις που ε, διατυπώνεται. Να ενισχυθεί λέγω, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή κατά την κατάρτιση της έκθεσης θα χρειαστεί να διευκρινίσετε το είπε και η πατή εκπρόσωπο, τι είναι αυτό, Ελεύθερε εκλογές, ελεύθερο τύπη, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, μεταρρύθμιση ε, της ασφάλεια, ισότητα ανδρών γυναικών, ε, δημοκρατικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων, ελευθερία του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε, όλα αυτά είναι οι άξονες και οι περισσυνοί. Και... Αυτή λοιπόν η βαθιά δημοκρατία που ορίζεται μέσα από όλους αυτούς τους στόχους θα πρέπει να είναι μια κατευθυντήρια γραμμή, ένα σειρμός που θα διαπερνά ε, όλους τους τομείς πολιτικής και συνεργασίας. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό άλλωστε είναι το θεμέλιο της αρχής περισσότερα για περισσότερα, το more for more. Ίσως αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε περισσότερο τι είναι αυτή η έννοια. Και μέσω του ιδίου του κανονισμού θα πρέπει να καλέσουμε όλα τα ενεχόμενα μέρη να το εκμεταλλευτούν, να το αξιοποιήσουν και να το υλοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι τα διακυβεύματα της οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας για να προχωρήσουμε σε μια ανάπτυξη του 21ου αιώνα. Όχι μόνο στην κοινωνική ένταξη, αλλά και με εξοικονόμηση ε, ε, των φυσικών πόρων και με χαμηλή παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ευκαιρία για μας να υποστηρίξουμε στη γειτονιά μας τέτοιου είδους οικονομίες ε, έτσι, με νυφαλιότητα και κάποια συγκράτηση στην ανάπτυξη. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα μπορούσα να προτείνω με λίγες τροπολογίες που θα κάνω στην έκθεσή σας. Γιατί γενικά συμφωνώ με την κατεύθυνση που δίδεται στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλότσο. Από την Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Μάγερς και ο Οδησίγητης. Ευχαριστώ τον κύριο Κούκαν για την έκθεσή του. Γνωρίζετε ότι η ομάδα μας έχει επικρίνει πολύ την πολιτική γειτονίας και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να είμαστε επικριτικοί διότι θα είμαστε και πιο απαιτητικοί. Καταρχήν διότι χρησιμοποιώντας την αρχή περισσότερα για περισσότερα more for more. Ε, δεδομένου ότι μιλούμε για γειτονικέ χώρες που κάνουν μεταρρυθμίσει αυτή τη στιγμή, αυτή η αρχή στη θεωρία είναι άψογη, όμως στην πράξη ε, α, παίρνοντας για παράδειγμα το πιο κοντινό το μοντέλο του Μαρόκου στο Μαρόκο έχει δοθεί ε, το ανώτερο καθεστώς εντός της πολιτικής γειτονίας το ε, το πιο ψηλό επίπεδο γειτονίας αυτή τη στιγμή έχει χορηγηθεί στο Μαρόκο σε ό,τι αφορά τις χώρες της Μεσογείου. Υπάρχουν συνάδελφοι που δίνουν το Μαρόκο ως παράδειγμα, αλλά αν ε, δούμε το, το δημοκρατικό επίπεδο του Μαρόκου, στην τελευταία, ε, στις τελευταίες εκλογές η συμμετοχή ήταν 23%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Αν το δούμε από πλευράς ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Μαρόκο ε, είναι αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει και κατέχει εν, μια αυτόνομη περιοχή ε, ε, που προσπαθεί να Ε, Συνεπώς θα πρέπει να εφαρμόσουμε καταρχήν την αρχή της ε, ανάγκης ε, της ε, κοινωνικής συνοχής. Δεύτερον, απασχόληση με θέση ποιότητας και τρίτον, βιωσιμότητα του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Η αρχή, περισσότερα για περισσότερα, δεν μας ικανοποιεί. Και έδωσε το παράδειγμα του Μαρόκου, αλλά θα μπορούσα να δώσω και, άλλο, και άλλα παραδείγματα, όπως το Ισραήλ που παρολίγο να του δώσουμε το ανώτερο καθεστώς. Ε, το οποίο έχει προς στιγμή ε, ανασταλεί αλλά ε, θα μπορούσε να δοθεί στο μέλλον. Θα μπορούσαμε και για το Ισραήλ να δούμε το κατά πόσον πληρεί τις αρχές και τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είμαστε επικριτικοί έναντι της ε, φιλοσοφίας του να προσπαθούμε η στρατηγική 2020 ε, ε, να επικρατήσει ως αρχή της πολιτικής γειτονίας. Δηλαδή να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σε αυτές τις χώρες το δικό μας καθρέφτο, το δικό μας είδωλο. Εμείς είμαστε εναντίον της στρατηγικής 2020 όπως είμαστε εναντίον της στρατηγικής Λισαβόνας. Είμαστε εναντίον του οικονομικού προσανατολισμού που ε, έχει την απελευθέρωση της αγοράς βασικό στοιχείο και χαρακτηριστικό της. Συνεπώ δεν θα μπορούσαμε να προβάλλουμε αυτέ τι πολιτικέ στι γειτονικέ χώρε, γιατί αυτή η οικονομική πολιτική έχει οδηγήσει στην καταστροφή το νότο τη Ευρώπη. Από την συνθήκη του Μάστρεχτ και μετά έχουμε μια δογματική προσέγγιση ε, που απαγορεύει την παρέμβαση στην οικονομία, ε, απαγορεύει την ύπαρξη ε, δημόσιων κρατικών εργαλείων παρέμβασης ε, που είναι εναντίον της ε, κρατικοποίησης συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας που είναι εναντίον του Δημόσιου Ταμείου Συνεπώς στην η ομάδα μου δεν πρόκειται να θέσει ως παράδειγμα για τις χώρες, τις γειτονικές χώρες κάτι το οποίο επικρίνουμε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί και πολύ πιο σαφείς. Και δύο ακόμα πραγματάκια. Πρέπει ε, να αναζητήσουμε ζώνες συνεργασίας και όχι ζώνες ελευθερής ελεύθερων ανταλλαγών. Για παράδειγμα, ε, η κυβέρνησή μου ανακοίνωσε μια σύμβαση με την Σαουδική Αραβία για την πώληση 250 τάγκς Αν αυτό είναι το παράδειγμα του περισσότερο για περισσότερα, τότε εμείς θα κατέβουμε από το τρένο. Ξέρετε, η Σαουδική Αραβία, έχουμε τη δυναστεία Σαούτ, στο ποινικό, στο ποινικό της κώδικα ε, έχει αντίθετα με τα δεδομένα των, του, των ε, Ηνωμένων Εθνών ε, τις ε, σωματικές ε, ποινές, δηλαδή ως ποινή, που δεν γίνονται εκλογέ κλπ. Και, και παρόλα αυτά εμείς τους πουλάμε 250 άρματα μάχης. Ο κύριος Κούκα λοιπόν θα καταλάβει ότι θα είμαστε πολύ επικριτικοί και απαιτητικοί σε σχέση με αυτή την καινούρια, τον καινούριο προσανατολισμό της πολιτικής γειτονίας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριο Μάγερ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο στην κυρία Υπρισάγια. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει διερμηνία από τα Σουηδικά. Ο κύριος Κούκαν μίλησε αγγλικά. Κάποιος πρέπει να μιλήσει σλοβάκικα και θα είμαι εγώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με το κείμενο του κυρίου Κούκαν. Είναι πάρα πολύ καλό και οι προτεραιότητες που μας ε, ανέφερε ο κύριος Κούκαν σήμερα εδώ είναι αυτές που με βρίσκουν και εμένα σύμφωνοι. Θα το διαβάσω το κείμενο πολύ προσεκτικά μια δεύτερη φορά και σε περίπτωση που έχω κάποιες ε, προτάσεις να κάνω θα τις αποστείλω στον κύριο Κούκαν υπό τη μορφή τροπολογιών. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να επεκτείνουμε το κείμενο περαιτέρω. Δεν θα πρέπει ούτε και να ε, το κάνουμε ένα κατάλογο με τις διάφορες επιθυμίες μας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιμένουμε όσο το δυνατόν πιο πιστοί στο πρωτότυπο. Ευχαριστώ πολύ και αν έχω κάποιες προτάσεις θα καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπυρσάγκητς και τώρα η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλους όσους εξέφρασαν την εκτίμησή τους ε, για το εν λόγω κείμενο. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω κάτι το οποίο μας δυσκολεύει ιδιαίτερα στη Φιλανδία. Μας ε, ανησυχεί ιδιαίτερα η μοίρα της βόρειας διάστασης ελοχεύει ο κίνδυνο να χαθεί αυτή η βόρεια διάσταση ε, όταν θα γίνει μεταφορά από την, ε, ε, στο μηχανισμό γειτονία και από την εταιρική σχέση γειτονία. Και νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση εδώ. Η βόρεια διάσταση δεν είναι σημαντική μόνο για τη Ρωσία, αλλά για όλη την περιοχή της Βαλτικής. Και είναι ζωτική σημασίας για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βαλτική θάλασσα. Αν το δούμε απλώς με όρους επιμελητείας είναι πολύ σημαντική για όλες τις βόρειες χώρες. Υπάρχει και η οπτική της Αρκτικής. Η βόρεια διάσταση λοιπόν είναι πολύ καλύτερο να παραμείνει στο μηχανισμό γειτονία και εκεί θα πρέπει να παραμείνει. Γνωρίζω ότι δεν ξέρετε όλοι ε, ποια είναι τα, ε, τα όσα περιλαμβάνει η Βόρεια Διάσταση, αλλά στο παρελθόν η Βόρεια Διάσταση κατέδειξε ότι μπορεί να συνεισφέρει ιδιαίτερα και να έχει απτά αποτελέσματα με πολύ ταπεινή χρηματοδότηση. Και φοβάμαι ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να μας οδηγήσει σε περικοπές στη χρηματοδότηση για τη βόρεια διάσταση. Για τη βόρεια όμως περιοχή της Ευρώπης αυτή η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να την συμπεριλάβουμε λοιπόν τη βόρεια διάσταση στο μηχανισμό εταιρική σχέση δεν θα επαρκεί για να καλύψει τι ανάγκε τη βόρεια διάσταση. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ αργό για να αλλάξει αυτή η κατάσταση λοιπόν, διότι ξέρω ότι στον όλο προγραμματισμό όλο αυτό μπορεί να φαίνεται ίσονο σημασία λεπτομέρεια, αλλά για μα στι βόρειε χώρε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακονσάρη. Πριν δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κορνάρο είναι εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Ε, good afternoon, Γεια σας, είμαι διευθυντής της σχέσης Ιτανίας ε, στην Κομισιόν. Ε, καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Κούκαν και για τη συνεργασία του μέχρι τώρα και από για, ε, ε, για πολλά από τα σχόλια που βλέπουμε στην έκθεση. Ε, ανέφερε την προσέγγιση πακέτου. Υπάρχουν κάποια σχόλια που αφορούν όλα τα ακτήματα του πακέτου, οπότε δεν πρόκειται να αναφερθώ σε οριζόντια θέματα όπως η κατεξουδότηση πράξη κλπ. Γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη σχολιαστεί. Ε, μας αρέσουν ιδιαίτερα ε, ορισμένα σημεία που ενισχύουν την πολιτική μας, για παράδειγμα η τροπολογία 30 για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στην γειτονιά. Ε, χαίρομαι που αυτό ενισχύει, ενισχύει την πρότασή μας. Ε, επίσης, είναι πολύ καλό το πόσο ο εισηγητής αντιλαμβάνεται την πρόθεση διαφοροποιημένης προσέγγισης. Για παράδειγμα, τροπολογία 42 είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και στο Συμβούλιο. Και εκεί, εκεί ελέγχθη ότι χρειάζεται πιο συγκεκριμένη γλώσσα. Δύο-τρία θέματα τώρα για τα οποία θεωρούμε πως οι προτάσεις είναι λίγο δύσκολο να ελοπιθούν. Πρώτον, τροπολογία 47 για, τα, για τον κοινό προγραμματισμό. Όλοι το υποστηρίζουμε, αλλά είναι δύσκολο στην πράξη αν υπάρχει απουσία συνεργασία από το κράτος ε, επίσης, τροπολογία 7, η ισορροπία ανάμεσα στις διαστάσεις, την ανατολική και την νότια διάσταση. Και αυτό είναι δύσκολο να το μεταφράσουμε σε γλώσσα σε ένα κανονισμό ε, και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε διαφοροποιημένη μας προσέγγιση. Ε, για το Ίδρυμα ε, το υποστηρίζουμε. Θέλουμε να εστιαστεί στην αρχή στην ε, γειτόνια, ε, όχι όμως να αποκλειστικά εκεί, ε, στην αρχή να εστιαστεί μόνο στο μηχανισμό γειτονίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βορειοδιάσταση, να καθισχάσω την συνάδελφο ότι μέσω της διασυνορικής ε, συνεργασίας σε αυτό το μέσο ε, έχουμε άνοιγμα και για την βόρεια διάσταση αλλά και άλλα μηχανισμοί όπως ε, τις εταιρικές σχέσεις ή οι τρεις θεματικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν την βόρεια διάσταση στο μέλλον. Συνεπώς δεν υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί στο περιθώριο. Αυτά τα λίγα δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ξανά ευχαριστώ τον εισηγητή για τις πολύ επικοδομητικές συζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον εκπρόσωπο της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Yes, good afternoon. It's Χαίρετε. Θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ε, για το μηχανισμό αυτό στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συμμετέχουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στις συζητήσεις άρα υποστηρίζω και υπογραμμίζω τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κ. Κορνάρο. Ευχαριστώ για τη συντομία σας και ε, τώρα ο συγητής μας ο κ. Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω εγώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Αρλάκη και την κυρία Φλότρο, συμφωνώ με τα όσα είπαν. Οι διευκρινήσεις που ανέφεραν ε, ότι θα κάνουν σε τροπολογίες είναι πάρα πολύ εύστοχες και συνδέονται ευθέω με τις δικές μου προθέσεις. Ε, ελπίζω να συνεργαστούμε για να το συμπεριλάβουμε στο μηχανισμό. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μάιερ, γνωρίζω τη θέση αυτή της πολιτικής σας ομάδας και μπορώ να συμφωνήσω με την πρώτη σας πρόταση ότι το ε, περισσότερα για περισσότερα είναι ε, αξιέπαινος αρχή αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Μα γι' αυτό άλλωστε προτείνουμε το συγκεκριμένο μηχανισμό και μέσο για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λαμπρό σχέδιο. Δεν θα αναφερθώ σε χώρες που μιλήσατε εσείς. Κοίταξε, η Σαουδική Αραβία δεν είναι μέλος της πολιτικής γειτονίας. Η κυρία Γιακονσάρη. Πρέπει να ξέρετε ότι συζητήσαμε το θέμα αυτό της ε, βορειοευρωπαϊκής διάστασης ε, θα το ξανασκεφτούμε. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τις ανησυχίες σας. Ε, φοβάστε μήπως παραγωνιστεί αυτή η διάσταση, δεν θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Το είπε όμως και ο κύριος Κορνάρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταλήξαμε και εμείς στο συμπέρασμα αυτό σε ό,τι αφορά τη Ρωσία. Συμπεριλαμβάνεται στο μέσο αυτό με το... Ε, κατάλληλο τρόπο η Ρωσία με τη διασυνοριακή συνεργασία και η συμμετοχή της ε, έχει διατυπωθεί με τρόπο σωστό, εύστοχο και αντικειμενικό. Ο κύριος Κορνάρο εξήγησε ότι η βόρεια ε, διάσταση μπορεί να ενταχθεί αλλού σε άλλα μέσα και σε άλλους μηχανισμούς. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός για τη γειτονία βασίζεται σε δύο εκθέσεις. Η μία ήταν του κυρίου Σίβιτς και η άλλη ήταν του Μάριο Ντάβιτ. Εσείς αναφέρατε και πολλά άλλα στοιχεία και την αρκτική διάσταση. Αν αρχίσουμε τώρα να προσθέτουμε διάφορα άλλα στοιχεία στο συγκεκριμένο μηχανισμό, φοβούμε ότι θα χάσει το στόχο του. Δεν θα βελτιωθεί, ούτε θα γίνει πιο ρεαλιστικός ο μηχανισμός. Πάντως κατανοώ ε, την ανησυχία σας για τη βόρεια διάσταση. Και τώρα, ε, σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Κορνάρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αναφέρθηκε σε διάφορες τροπολογίες. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Προφανώς και είναι δύσκολα και περίπλοκα αυτά τα ζητήματα, αλλά αν χρησιμοποιήσουμε τη θετική προσέγγιση που μέχρι τώρα επέδειξαν σχεδόν όλοι, ε, θα καταλήξουμε σε ένα αποδεκτό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, όλοι, Πρόεδρος. Τελειώνει εδώ η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Οχτώ επιτροπές γνωμοδοτούν για την έκθεση αυτή για το μηχανισμό γειτονίας. Περνούμε στο επόμενο θέμα της απογευματινής μας ημερησίας διάταξης. Πρώτη αντιλαγή απόψεων για νομοθετική έκθεση σχετικά με το μέσο ε, συνεργασία με τρίτε χώρε, Συγητή είναι ο κύριος Μάριο Μάουρο. Θα ήθελα να σα θυμίσω όμως ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου συμμετέχει βάσει του άρθρου 50 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινοβουλίου για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο και την οικονομική συνεργασία. Εκεί η συντάκτρια γνωμοδότηση είναι η κυρία Αντρικέινε. Στις 7 Ιουνίου θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση κατά τη διάρκεια τη συνεδρία τη Επιτροπή μα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μάουρο, για να μα παρουσιάσει την έκθεση του. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και ομολογώ ότι θα ήθελα να διασταυρώσω λίγο απόψεις ε, με τους σκιώδεις εισηγητές σε αυτή την προπαρασκευαστική ε, διαδικασία πριν κάνω την πρόταση κειμένου μου και να δω και τις γνωμοδοτήσεις των υπολείπων επιτροπών. Περίμενα όμως και τις αποφάσεις της διάσκεψης των Προέδρων και της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών για την ε, νομική γνωμοδότηση που καθόρισε ποιος έχει αρμοδιότητα μεταξύ ΜΟΝ και της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου και ελπίζω ότι πλέον ε, επειδή καθορίστηκε και ποιο ανού είναι η αρμοδιότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μπορέσω να συνεργαστώ και με την κυρία Αρντρικέινε και με τους κοιόδησης εισηγητές. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, για το μέσο εταιρικής σχέσης ε, είναι πολυπίκυλη. Εγώ στάθηκα σε τρία σημεία και σε αυτά έχω επικεντρώσει και τις τροπολογίες που κάνω. Καταρχάς το θέμα των χωρών δικαιούχων αυτών των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτωθούν από το Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε πόσο ευρεία μπορεί να είναι ε, η συμμετοχή των διαφόρων χωρών και ε, τα σημαντικά ζητήματα που θα καθορίσουμε για το μέσο αυτό και επίσης ε, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω αυτού του μηχανισμού εταιρικής σχέσης. Όπως είπε και ο συνάδελφος Κούκαν, δεν θα σχολιάσω και εγώ εδώ το θέμα των κατεξουσιοδότης συμπράξεων, διότι ο κύριος Μπρόκ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό σήμερα το πρωί και όπως γνωρίζουμε όλοι συμφωνούμε με τις θέσεις του. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένας δημοκρατικός έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το στρατηγικό προγραμματισμό για το κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και αυτό είναι υψής της σημασίας, γι' αυτό και ε, το ίδιο ισχύει και για το μηχανισμό εταιρική σχέσης και βρίσκεται σε αυτό το κοινό μας όραμα. Όσον αφορά τώρα τις χώρες δικαιούχους ε, για αυτά τα προγράμματα συνεργασίας που χρηματοδετούνται από το μέσο εταιρικής σχέσης, εγώ ε, θέλησα να ενισχύσω τον παγκόσμιο χαρακτήρα αυτού του μέσου. Δηλαδή, το μέσο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο με βάση τους στρατηγικούς εταίρους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για όλες τις τρίτες χώρες που είναι στρατηγική σημασία για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στρατηγικό στοιχείο λοιπόν, κατά την άποψή μου, δεν καθορίζεται από τη χώρα αυτή καθ' αλλά από το συμφέρον που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις σχέσεις της με μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Ε, θα πω δύο λόγια παραπάνω για το σημείο αυτό, διότι θεωρώ ότι είναι η πλέον κατάλληλη προσέγγιση για να εξηγήσουμε ότι αυτό το μέσο ε, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τα ίδια κονδύλια με τα υπόλοιπα μέσα, έχει αρκετές δυνατότητες ευελιξίες και αυτό σημαίνει ότι το κατατάσσουμε στην κατηγορία των πολύ χρήσιμων μέσων, διότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στρατηγικές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντική, διότι θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι μόνο για τις χώρες που ήδη διαθέτουν ε, καθεστώς ε, στρατηγικού εταίρου, αλλά και για όλες τις χώρες που είναι σημαντικές και σε γεωγραφικό αλλά και σε θεματικό επίπεδο για τα συμφέροντα τα οποία σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρήσει ότι είναι καθοριστικές σημασίες για το μέλλον της. Όσον αφορά τώρα τη μέθοδο, εγώ πρότεινα κάποιες τροπολογίες ε, που όπως και ο κύριος Κούκαν επισημαίνουν τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στιών ε, καθορισμό αυτών των προγραμμάτων συνεργασίας με τρίτες χώρες. Πρέπει να πω ότι εδώ με υποστηρίζουν Συγγνώμη, τη θέση μου την ε, ε, έχω στηρίξει στη πείρα που έχω αποκτήσει στα 13 χρόνια που είμαι εδώ ως Ευρωβουλευτής ε, και την εμπειρία που έχω από χώρες οι οποίες είχαν κυβερνήσεις που κατόπιν έγιναν καθεστώτα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε το σημείο αυτό και επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει μια πολύ αυστηρή ερωσιμότητα εδώ θα πρέπει να δημιουργούμε μηχανισμούς που θα μας επιτρέπουν να αναστείλουμε τα προγράμματα συνεργασίας το οποίο θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα μοχλό πίεση για να προωθήσει τις αρχές της. Για παράδειγμα, το σεβασμό κάποιων θεμελωδών αρχών. Ε, νομίζω ότι το ανέφεραν και αρκετοί συνάδελφοι στην προηγούμενη συζήτηση. Όλες εκείνες τις πτυχές ε, που δεν θα πρέπει να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συγκεκριμένε διεκδικήσει και να βλέπει τα πάντα ω ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να θέτει συγκεκριμένου όρου. Και πέρα από αυτέ τι θεμελιώδει αξίε, θα πρέπει να προασπίζει και τα συμφέροντά τη. Όπω για παράδειγμα, ε, να φροντίζει τι επενδύσει τη ε, σε τρίτε χώρε. Τέλο, όσον αφορά του τομεί συνεργασία, και αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό, το οποίο καθορίζει και την ίδια την ουσία αυτού του μέσου εταιρική σχέσης. Οι προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παράρτημα, κατά την άποψή μου, καταδεικνύουν ότι αυτή το μέσο εταιρική σχέση είναι κατά βάση εξωτερική πολιτική. Αλλά ίσω είναι πάρα πολύ γενικόλογοι τα όσα λέγονται στο παράρτημα και ελοχεύει ο κίνδυνο να χαθεί αυτή η εξωτερική διάσταση του μέσου και κάνω συγκεκριμένε τροπολογίε, ώστε να αναφέρεται σαφώ αυτή η πολιτική εξωτερική διάσταση του μέσου εταιρική σχέση. και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον διμερή και πολυμερή διάλογο, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο την παγκόσμια διακυβέρνηση και πρωτίστως να δώσουμε τους πόρους για να διευκολύνουμε την εφαρμογή των συμπερασμάτων ε, διεθνών ε, ε, επικεφαλής, όπως για παράδειγμα τα όσα καθορίζει το G20, και από εκεί και πέρα να σταθεροποιήσουμε τις αξίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα στη σχέση μας με αυτούς τους εταίρους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους για την ε, προσοχή τους και είμαι εν αναμονή των παρατηρήσεων και των επικρίσεών τους. μικρόφωνο, Oh, <laughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάουρο για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αντρικέιν. Thank you, Mr. Chairman. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι χτες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έγινε μια ανταλλαγή απόψεων για τις ε, τροπολογίες επί του προσχεδίου κανονισμού για αυτό το μηχανισμό. Και νωρίτερα σήμερα το είπε και ο κύριος Μάουρο, ε, έλαβε χώρα μια πολύ χρήσιμη συνάντηση μαζί του για να διευκρινίσουμε τα πράγματα και να καταλάβουμε καλύτερα τις, να γίνουν πιο καλά κατανοητές τροπολογίες. Το, ο μηχανισμός εταιρική σχέση είναι μία, ένα από τα εργαλεία εξωτερικών, εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υποστηρίζει την πολιτική εξωτερική, την ε, εξωτερικών σχέσεων. Έτσι που διαβάζουμε εμείς το κείμενο, έχει τρεις στόχους. Πρώτον, να εφαρμόζει την διεθνή διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεύτερον, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή των Εμπορίου, να βελτιώσει την πρόσβαση σε αγορές και να αναπτύξει το εμπόριο, τι επενδύσει ε, και να δημιουργήσει καινούργιε επιχειρηματικέ ευκαιρίε για τι ε, κυρίω μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, να βελτιώσει την ορατότητα και την κατανόηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσει τα συμφέροντα και τι αρχέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. η Επιτροπή ΙΝΤΑ ιδιαίτερω ενδιαφέρεται για το δεύτερο από αυτού του στόχου, όπω σα είπα. Σύμφωνα με αυτούς τους ε, στόχους έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις πτυχές διεθνούς εμπορίου. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για να υποστηριχθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα και να συνεισφέρει στην μείωση του κινδύνου προστατευτισμού, να προωθήσει τις κοινωτικές αρχές και να δημιουργήσει καινούργιες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχουμε εκπροσώπους της ε, Κομισιόν εδώ πέρα και της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λόγο θα ήθελα να τους ζητήσω τη γνώμη τους ε, για την τροπολογία που έχουμε υποβάλει και είναι σημαντική για τις δύο τροπές. Είναι η τροπολογία που, της ίντα που προτείνει να μειωθεί το μερίδιο των ε, μη σημαντικών ε, διαφοροποιήσεων του προγράμματος από το 20% στο 10%. Η τροπολογία υποβλήθηκε από τον Μάριο Μάουρο. Προτείνει την διαγραφή της παραγραφού. Εμείς προτείνουμε την μείωση ε, από το 20% στο 10%. Η Κομισιόν θέλει να διατηρήσει το μερίδιο αυτό στο 20% αλλά είναι πολύ ψηλό. και ε, στο ε, τα πολιετή ενδεικτικά προγράμματα που περιέχουν ε, τις προτεραιότητες μας μπορεί να φυγούν από αυτό το ποσοστό. Είναι πολύ σημαντικό και υποστηρίζω την θέση του εισηγητή της ΑΦΕΤ ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί το πεδίο αυτού του μηχανισμού, αυτού του κανονισμού μόνο στις μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, νομές πολιτείες και που είναι μεγάλοι σημαντικοί παίκτες αλλά να περιλάβουμε και άλλες περιοχές και χώρες ε, καθώς επίσης και εδάφη που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντα από στρατηγική πλευράς για πολιτικούς και οικονομικούς εμπορικούς ε, λόγους. Υποστηρίζω τις τροπολογίες του Μάριο Μάουρο για αυτό το θέμα. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ανδρικίνη. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης. Είναι κοινή ομάδα, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο. Κύριος Ματιέ από την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζω ότι είμαστε μια κοινή ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το μέσο εταιρικής σχέσης. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια γενικά σχόλια, αλλά προσαρμοσμένα στις ειδικέ ερωτήσεις που κάνατε. Βεβαίω θεωρούμε εμείς ότι το μέσο εταιρικής σχέσης που προτείνουμε έχει ένα στοιχείο καινοτόμο, που είναι η παγκόσμια εμβέλειά του, το τονίσατε και εσείς στις τροπολογίες που κάνετε και του εισηγητού είναι σε αντίθεση με το ICI και το ICI Plus που είχαν περιορισμένο γεωγραφικά πεδίο εφαρμογής. Εδώ υποστηρίζουμε την εξωτερική ε, διάσταση της πολιτικής μας και της ε, στρατηγικής του 2020. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, ε, η ενεργειακή ασφάλεια. Τονίζουμε πολύ και ενισχύουμε αυτούς τους στόχους. Αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι στο μέσο αυτό προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την αντίληψη της αναπτυξιακής. Δεν υπάρχουν απαιτήσει ODA ε, για χώρες που ε, αναπτύσσονται και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίω. Δηλαδή έρχεται να καλύψει ένα κενό το μέσο εταιρικής σε σχέση με τα όσα έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας στον τίτλο 4 θα επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με χώρες στρατηγικές για τα συμφέροντά της, να υποστηρίξει διαλόγους πολιτικής. Αυτό αφορά εντός εισαγωγικών επίσημου στρατηγικούς εταίρους αλλά και άλλες χώρες που δεν μπαίνουν στον επίσημο ορισμό του στρατηγικού μας εταίρου. Το είπε και ο εισηγητής είναι και σημαντικό για την Ένωση να αναπτύξει εταιρική σχέση με χώρες που δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει, είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, αλλά και η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία. Κατά τα άλλα είναι χώρες με τις οποίες ήδη έχουμε ε, βαθιά ε, συνεργασία με προγράμματα δράσης, με συμπεράσματα συνόδων κορυφή. Μερικέ φορέ έχουμε και συμφωνίε, πλαίσιο, αλλά γενικά Είμαστε σε μια διαδικασία ενημέρωσης και των εμπορικών μας συμφωνιών αλλά και των συμβατικών μας σχέσεων με ένα ενημερωμένο και πιο επίκαιρο πλαίσιο πλέον. Βλέπω στροπολογίες σας θέματα που σταχειολόγησα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ε, παγκόσμια δεκυβέρνηση ή ε, από την ατζέντα του G20, η συμμετοχή και συνεργασία ε, της κοινωνίας των πολιτών και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και για χώρες μέσου εισοδήματος που έχουν ξεφύγει από τη διμερή σχέση αναπτυξιακής βοήθειας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Να θυμίσω μόνο ότι για τις χώρες μέσου εισοδήματο ε, μπορούν ε, επιμέρους και κατά καιρού να χρηματοδοτούνται και από το μέσο της αναπτυξιακής βοήθειας, το DCI, σε διάφορα θέματα. Επίσης αναφερθήκατε και στη ρήτρα αναστολής. Σας διαβεβαιώ ότι το συζητά αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο. Και αν μου επιτρέπετε να μιλήσει και ο συνάδελφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποια ζητήματα συγκεκριμένα εφαρμογής και υλοποίησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά στοιχεία μόνο. Σε σχέση με το ποιοι θα κληθούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο μέσο. Ε, ε, λίγες παρατηρήσεις σε σχέση με τις τροπολογίες. Αυτή είναι του δικαιούχου αναφέρεται σε ορισμένες ε, περιπτώσεις και ε, στις αιτιολογικές σκέψεις αλλά και στο διατακτικό και στα άρθρα δηλαδή. Όταν μιλάμε για όφελο, αν είναι αμοιβαίο όφελο ή όφελο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν ξέρω, μπορεί να οδηγήσει αυτό σε παρερμηνίες και παρεξηγήσει για τι χώρε δικαιούχου στα αγγλικά beneficiary countries, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο. Ε, γενικά μια παρατήρηση για τους δείκτες. Σε διάφορα σημεία των τροπολογιών και πάλι χρησιμοποιείται αυτή η διατύπωση περί δικτών. Αυτό το μέσο θα πρέπει να ε, χρηματοδοτεί έργα που να πιάνουν το από τα χρήματα και να υπάρχει και λογοδοσία. Αλλά τι θα πει τώρα εξάντε ορισμός εκ των προτέρων, ε, καθορισμός συγκεκριμένων ε, ωφελιών για τις δικαιούχες χώρες. Και είναι πολύ δύσκολο εκ των προτέρων να εκτιμήσει κανείς ποιο όφελος θα έχει ε, αυτό το μέσο ως υποστηρικτικό της διπλωματικής μας προσπάθειας και συνεργασίας με τις χώρες αυτές. Χρειάζεται λίγη προσοχή γιατί όταν μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες είναι και πάρα πολύ ε, καθοδηγητική, περιγραφική διατύπωση, γιατί δεν είμαστε αρκετά ευέλικτοι ούτε αρκετά ευθυγραμμισμένοι με την πραγματικότητα σε αυτή την περίπτωση. Καλό θα ήταν λοιπόν στα έγγραφα προγραμματισμού να αναφέρεται κάτι τέτοιο που αλλάζουν και πιο εύκολα από ότι ο ίδιος ο κανονισμός. Αυτό ήταν μάλλον ένα γενικότερο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τα σχόλιά σας και για να ολοκληρώσει τη συζήτηση και να συνοψίσει παρακαλώ και πάλι ο συγητής ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από αυτά που άκουσα, κατανοώ πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας την κυρία Αντρικέινε, με την οποία είμαι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε μια πραγματική συνεργασία, δηλαδή να συμφωνήσουμε επί των περισσότερων θεμάτων, τώρα που ξεπεράστηκε και το ποια η ε, Επιτροπή είναι αρμόδια επί της ουσίας για το ζήτημα. Να ευχαριστήσω και την κυρία Αντρικίνη και για έναν ακόμα λόγο, διότι δικαίως έθεσε το θέμα αυτό του μηχανισμού σε ε, ποσοστό. Εγώ ήθελα ένα 10% αλλά ακούγοντας τις παρεμβάσεις της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δικαίως το ζητά αυτό το 10% διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση να μας δώσει κάποιο συγκεκριμένες ε, πληροφορίες και ε, είδα ότι δεν μου απάντησε κανείς το ερωτηματικό της κυρίας Αντρικέινε. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης διότι διευκρίνησε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μηχανισμός και πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει ευέλικτος και να είναι ένα μέσο στρατηγικού προσανατολισμού. Ευχαριστώ επίσης ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις παρατηρήσεις του, διότι ήταν αυτός που με έκανε να καταλάβω περισσότερο από όλους ότι με τις τροπολογίες μας έχουμε επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα θέματα. Να εξηγηθώ. Πολλές φορές ε, μας λένε πολλές λεπτομέρειες όταν ε, έχεις βάλει κάτι που ενοχλεί, όταν έχεις συμπεριλάβει κάποια στοιχεία τα οποία χτυπούν φλέβα και ε, νομίζω ότι όπως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και θα δούμε τι παρατηρήσεις θα γίνονται, θα δούμε τι είναι αυτό που δημιουργεί τόσο σοβαρό πρόβλημα στην Επιτροπή. Διότι εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά ε, τους δικαιούχους ε, και όσον αφορά και τους ε, εκ των προτέρων ε, καθορισμό των δικαιούχων. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να καθορίσουμε μία σχέση με τρίτες χώρες, τις οποίες δεν χρειάζεται πλέον να συνδράμουμε ή μπορεί και να πρέπει να τις συνδράμουμε, αλλά στη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχουν μία στρατηγική σημασία ιδιαιτερότητα, που είναι στρατηγική όχι μόνο για τη δική τους εξέλιξη ή για τη σχέση που καθορίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τους στόχους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από στρατηγική σκοπιά. Σας ευχαριστώ όλους, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είμαι βέβαιο ότι θα συναντηθούμε και θα συνεχίσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων πριν ε, την κατάθεση τροπολογιών και επομένως ε, φαντάζομαι ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι ακόμα πιο χρήσιμη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάουρο. Και με αυτό ολοκληρώσαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 14η Ιουνίου. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο ζήτημα, αλλά επειδή δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Βιγγένη, ο εισηγητής, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε πέντε λεπτά και ελπίζουμε ότι ο κύριος Βιγγένη θα είναι εδώ. Gonzato, potrebbe sostituire lei Θα μπορούσατε να αντικαταστήσετε εσείς τον κύριο Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με το μέσο προενταξιακής βοήθειας, το σημείο 10. Ήρθε ο συνάδελφος Βιγγένιν, καλώς ορίσατε. Ο οποίος είναι εισηγητής ε, για το κείμενο αυτό. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης για το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας. Ο κύριος Βιγγένιν έχει προτείνει αρκετέ τροπολογίε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βελτιώσει τη μελλοντική χρηματοδότηση της διαδικασίας διεύρυνσης και να κάνει τη διαδικασία πιο διαφανή, πιο αποτελεσματική και συνεκτική με του στόχου τη διεύρυνση. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βιγγένιν, Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κορνέλισεν. Πριν από τον εισηγητή, γιατί το έχει ζητήσει, έχει κάποιο λόγο η κυρία Κορνέλισεν, αν συμφωνεί βέβαια και ο εισηγητής. Συμφωνείτε κύριε Βιγγένιν. Δύο-τρία λεπτά, η κυρία Κορνέλισεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Πρέπει να φύγω γιατί συνεδριάζουν συντονιστές σε άλλη επιτροπή. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον εισηγητή. Δεν θα παραμείνω για τις απαντήσεις, αλλά είναι βοηθή μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική του εργασία. Ήδη είχαμε συζητήσει για το θέμα του, γιατί εγώ είμαι συντάκτρια γνωμοδότης Επιτροπής Απασχόλησης. Καλωσορίζω τις προτάσεις το εισηγητού για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, προβολή, δημοκρατία κτλ. Συμφωνώ με τα περισσότερα. Έχω μερικές ερωτήσεις. Το ένα έχει να κάνει με το 5% που θα μπαίνει σε ένα αποθεματικό για να επιβραβεύει τις καλές επιδόσεις. Καταρχήν είναι καλή ιδέα, αλλά με ενοχλεί λίγο το γεγονός ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του προενταξιακού μέσου σήμερα είναι να ε, απορροφώνται, να απαντώνονται καν τα κονδύλια με το σωστό τρόπο. Ορισμένες χώρες δεν έχουν απορροφήσει το 12 κονδύλια του 2007. Δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο αυτό εργαλείο για να προωθήσουμε και να δημιουργήσουμε ε, καλές συμπεριφορές. Ε, αυτή είναι η άποψή μου. Θα ήθελα και την άποψη του εισηγητού. Δεύτερον, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε τι προσπαθείτε ακριβώς να κάνετε με τις τροπολογίες 12 και 13 για τις κάτι εξουσιοδότηση πράξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη μία τροπολογία το αναδιατεπώνετε και στη δεύτερη το αφαιρείτε. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε. Και τρίτον, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε πώς θα οριστούν ακριβώς οι στόχοι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στην εκπόνηση του κοινού στρατηγικού πλαισίου και ε, των εγγράφων για την κάθε χώρα ξεχωριστά των στρατηγικών. Και πάλι σε μια τροπολογία το αναδιατυπώνεται και σε μια άλλη τη 15 το διαγράφεται τελείως. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Πώς το φαντάζεστε, σίγουρα μπορεί να είναι καλή, αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει. Επίσης, ε, εγώ παλεύω ακόμα με ένα πρόβλημα. Πώς θα γίνει με την απορρόφηση των κονδυλίων να ε, πηγαίνουν και να κατευθύνονται στις σωστές ε, κατευθύνσεις, να καταπολεπούμε την απάτη. Δεν έχω εγώ καμία πανάκια ή μια θαυμαστή ιδέα να προτείνω. Θα ήθελα τα σχόλιά σας. Και τέλος, χαίρομαι πολύ που πολλές από τις ε, προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης ε, έχουν υιοθετηθεί από τον κύριο Βίκιν. Ελπίζω να τον ε, πίσω στους συμβιβασμούς να δεχτεί και άλλες από τις προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και προσβλέπω στη συζήτηση για το μέσο πρωταξιακής βοήθειας. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στον συγητή, τον κύριο Βιγγένιν. Έχετε το λόγο. Πόσο χρόνο μου δίνετε, Πρόεδρε. Οκτώ με δέκα λεπτά. Και δύο δώρο για μένα, από μένα. Ε, ορισμένες από τις απαντήσεις θα τις ε, βρει, βρει η κυρία Κορνέλη στην απάντησή μου, ε, στην ομιλία μου. Δεν θα σας ε, παρουσιάσω το, τον ίδιο το μηχανισμό ε, πρενταξιακής βοήθειας ε, των IPA. Νομίζω πως λίγος πολύ ξέρετε τι είναι και ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρει. Να πω όμως ότι μέσω αυτού του ανανεωμένου μηχανισμού η Κομισιόν έλαβε ήδη στην αρχή της πρόταση υπόψη ορισμένες από τις αδυναμίες του προηγούμενου μηχανισμού, της πρώτης εκδοχής του IPA. Προτείνει λοιπόν ένα πιο ευέλικτο μηχανισμό με πρόσβαση που δεν συνδυάζεται πια με το καθεστώς αν είναι υποψήφια ή ενδεχόμενη υποψήφια χώρα η δικαίωχος χώρα. Το σημαντικό είναι οι δυνατότητες που έχει η συγκεκριμένη χώρα να υλοποιήσει τα προγράμματα και να απορροφήσει τα ποσά. Είναι δηλαδή πολύ πιο εύχριστος αυτός ο καινούργιος μηχανισμός. Η απορροφητικότητα των κοντιλίων του μηχανισμού επίσης θα είναι πιο εύκολη για τις δικαιούχες χώρες, αλλά είναι και πιο στρατηγικά στοχευμένος. Προτείνει ε, την αναεξάμεινο εξέταση των προγραμμάτων, αντί την ετήσια εξέταση κομισιών, ε, Επίσης θέτει και συγκεκριμένους όρους, ε, προϋποθέσεις, για παράδειγμα βελτίωση της ε, διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών. Ο μηχανισμός αυτό σίγουρα είναι καλύτερο από ότι ο προηγούμενο, η προηγούμενη εκδοχή του. Πριν περάσω σε συγκεκριμένες προτάσεις, να πω ότι στην διαδικασία της ε, προετοιμασίας των τροπολογιών μας, ε, ήρθαμε σε επαφή με ένα αριθμό ενδιαφερομένων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις δικαιούχες χώρες διοργανώσαμε μια πολύ επιτυχή κατά την άποψή μου ακρόαση και λάβουμε υπόψη τις ε, απόψεις που ακούστηκαν στις προτάσεις μας. Η κυρία Κορνέλιεσεν το είπε ήδη, αλλά να πω κι εγώ ότι έκανα ό,τι μπορούσα να ενσωματώσω τις ε, προτάσεις, ε, στις προτάσεις τις περισσότερες ιδέες και απόψεις των διαφόρων επιτροπών. που εξέδωσαν γνωμοδοτήσεις. Προς το παρόν δεν έχω καταφέρει να τα λάβω όλα υπόψη, ε, να τα συμπεριλάβω όλα, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία διαφωνώ. Οι προτάσεις οι οποίες δεν συμπεριλήφθησαν στις τροπολογίες έχουν περισσότερο σχέση με το γεγονό ότι πηγαίνουν πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ ειδικέ και παρόλο ότι θα ήθελα και εγώ προσωπικά και το Κοινοβούλιο ο μηχανισμός να γίνει πιο σαφής, πιο ειδικό. Δεν πρέπει να ε, πάμε και υπερβολικά μακριά, πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία. Η πρόκληση ήταν να εξασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα σε πολύ στο ειδικό και στο γενικό. Δεν θέλουμε ε, να είμαστε πολύ γενικοί για να μην ε, χάσουμε την διαφάνεια, ε, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε και πάρα πολύ ειδικοί, εξειδικευμένοι. Να πω δύο λόγια για τις βασικές προτάσεις μας. Καταρχήν, ε, κατεξιοδότηση πράξης είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στον, ε, στην μηχανισμό της, ε, στον κανονισμό της κοινή προσέγγισης. Ε, προτείνεται ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξοδοτήσουν την Κομισιόν να προετοιμάζει τα στρατηγικά, τα έγγραφα στρατηγικών προγραμμάτων με, τις, ε, με τους γενικούς στόχους, προτεραιότητες, προτεραιότητες κλπ. και να τα υιοθετεί ως κατεξοδότηση πράξη για να εξασφαλίσουμε ε, ε, ε ελαστικότητα αλλά χωρίς να χάσουμε τις βασικές μας αρχές. τα στρατηγικά προγράμματα, τα στρατηγικά έγγραφα, για παράδειγμα, θα υιοθετούνται ως κατεξοδότηση πράξη αν με το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κοινή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, όλα, για όλους τους μηχανισμούς. Και ελπίζω να βρεθεί μια λύση. Μετά, για το πεδίο εφαρμογή ε, της, ε, περιοχής, ε, της διάφορες πολιτικές, ε, δεν ήταν σαφή θέση στο πεδίο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αλλάξει λίγο τις ε, πολιτικές, τις περιοχές πολιτικής. Ε, έχουμε ενημερώσει λίγο ορισμένες υποπαραγράφους. Θα δείτε στην πρότασή μας αυτές τις τροποποίησεις. Η αιτιολογική ε, έκθεση του κανονισμού αναφέρεται επίσης στην απόδοση ε, η Κομισιόν δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα ε, και δεν έχουν συμπεριληφθεί καθόλου διατάξει τον κανονισμό για αυτό το θέμα. Εγώ προτείνω να προσθεθούν το άρθρο 1, καινούριο άρθρο 13α, μέχρι 5% του συνολικού ποσού να ε, ε, μπαίνει σε ένα αποθεματικό για να επιβραβεύει αυτούς που έχουν τις καλύτερες αποδόσεις. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για να λάβουμε πραγματικά υπόψη την απόδοση. Να επιβραδεύουμε αυτούς που έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα με τις μεταρρυθμίσεις. Θα μπορούσαμε να, να αυξάνουμε ε, τη χρηματοδότησή τους. Αυτό δεν έχει σχέση, απαντώντας στην κυρία Κορνέλιος, Κορνέλισεν, ε, δεν, ε, δεν, είναι... δεν αποτελεί μια προσπάθεια να ε, δαπανίσουμε περισσότερα κονδύλια. Θέλουμε αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις να επιβραβεύονται. Όπως είπα, επίσης αυτό θα πρέπει να γίνεται με πολύ σαφή κριτήρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του κανονισμού, αλλά μέσω του κοινού στρατηγικού πλαισίου, με του κοινού πλαισίου στρατηγικής. Η διασυνορική συνεργασία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με μεγαλύτερα κονδύλια σύμφωνα με την πρόταση Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επιτροπής Ρέτζι. Προτείνουμε να αυξηθεί το ποσοστό της διασυνοριακής συνεργασίας από το 3% στο 7%. Μέχρι 7%. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι 7%. Πρέπει να δούμε και αν οι δικαιούχες ε, χώρες ε, έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης. Επίσης αυτή η διασυνορική συνεργασία θα προετοιμάσει αυτές τις ε, χώρες για ένταξη γιατί θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις γνώσεις των κρατών, της Ευρωπαϊκής, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τις χρησιμοποιήσουν όταν ενταχθούν. Είναι σημαντικό επίσης να διευκρινιστεί, ε, να διευκρινιστούν τα του άρθρου 2, ε, δείκτες ε, πρόοδου, οι οποίοι αναφέρονται στα έγγραφα προγραμματισμού. Θα πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα και το κείμενο του κανονισμού θα πρέπει να, να δίνει σαφή αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για τη χρηματοδότηση και να καθορίζει τους δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την ε, επιβεβαίωση και τη μέτρηση της πρόοδου. Θέλουμε να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η δυνατότητά της να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο, ε, σε διάφορες φάσεις του κύκλου χρηματοδότησης. Θέλουμε να διευρύνουμε λίγο τους γενικούς στόχους της, ε, του μηχανισμού ε, όχι μόνο την τήρηση, την πλήρωση των ε, ε, κριτηρίων εισόδου, θα πρέπει να βελτιωθεί η σταθερότητα και η ευημερία. Δηλαδή ο μηχανισμός να βοηθάει στη βελτίωση της σταθερότητας και της ευημερίας, καθώς επίσης και της ανάπτυξης της δικαιούχες χώρες. Ε, επίσης έχουμε περιλάβει τις καλές σχέσεις γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία στους ειδικούς στόχους του άρθρου 2, επίσης ε, την κοινωνική εσωμάτωση των προσφύγων και των εκτοπιστέντων. Αυτό αφορά κυρίως την, τα Δυτικά Βαλκάνια, όχι την Ισλανδία τόσο πολύ. Ε, προτείνουμε επίσης και κάποιες αλλαγές σε σχέση για να, μάλλον για να ε, χρησιμοποιήσουμε ε, τη διατύπωση της συνθήκης για να είμαστε έτσι συνεπείς σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Τέλος, η κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται με βάση τις επιτυχίες τη και την απόδοσή της. Ε, αυτό είναι η ιδιωτική σκέψη παρθμών 5 συγκεκριμένα. Και επίσης λέμε σε συνεργασία με άλλους δωρητές, συμπεριλαμβανομένε και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Μιλάμε επίσης για τα κοινωνικά θέματα, κοινωνική ένταξη, τα ε, κινητικότητα του... των εργαζομένων, μειοψηφ... κλπ. Ένταξη των μειονοτήτων κλπ. Ε, τέλος, θέλουμε να ενισχυθεί η παρουσία, η ορατότητα του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το θέμα αυτό το συζητήσαμε και σε σχέση με άλλους μηχανισμούς. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν πρέπει κάτι παραπάνω να κάνει για να γίνουν πιο ορατά τα αποτελέσματα και η ίδια βοήθεια. Όχι μόνο στις δικαιούχες χώρες, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που μας βοήθησε στην προετοιμασία της έκθεσής μου. Ε, ήταν πάντοτε διαθέσιμη. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα είναι στο πλευρό της Κομισιόν. Έχουμε κοινούς στόχους, κοινέ προτεραιότητες και πιστεύουμε ότι από κοινού, Κομισιόν και Κοινοβούλιο μπορούμε να πετύχουμε πιο πολλά για το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας γνωρίζοντας και τις συζητήσεις στο Συμβούλιο για αυτό το μηχανισμό, θεωρώ πως δεν θα παρουσιαστούν σοβαρά, ανεπίλητα προβλήματα στις, ε, σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Υπό την προπόθεση θα λυθεί το θέμα των κατεξουδότηση πράξεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος, η κυρία Νέμσκη, η Οδύση Συγήτρια. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Βιγγένινγκ ε, για τα όσα έκανε στο σχέδιο έκθεση για την πρόταση για αυτό το μηχανισμό προενταξιακή βοήθεια. Νομίζω ότι αντιμετώπισε πολλέ από τι ελλείψει αυτού του ε, κανονισμού και ε, μα δίνει και κατάλληλε κατευθύνσει για τα όσα θα κάνουμε εμείς στην Επιτροπή μα. Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης Επιτροπής Προϋπολογισμών θα ήθελα να επικεντρωθούμε περισσότερο στους στόχους ε, της βοήθειας και τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνουν οι χώρες δικαιούχοι. με ενδιαφέρει ε, το τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή ε, χρηματοδότηση, να γίνεται σωστό υπολογισμό ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψει και να διασφαλίζεται ότι δεν κατασπαταλώνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογωμένων ιδίω εν καιρό Επιπλέον, όπως ε, και ε, μετά όσα συζητήσαμε για τον κοινό εφαρμοστικό κανονισμό σήμερα το πρωί, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική διεύνηση. Βλέπω ότι ο κύριος Βιγγένιν έχει λάβει υπόψη κάποιες από τις συστάσεις μου στο σχέδιο έκθεσής τους. Ως κυριώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα εξετάσω κάποια από τα εξή θέματα. Καταρχάς, θα εξετάσω περαιτέρω τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού απόδοσης, ε, το οποίο υποστηρίζω και εγώ και θα ήθελα να ε, έχει ένα 5% της χρηματοδότησης εγγυημένο. Δεύτερον, θα δω ε, περαιτέρω το κύκλο ζωής των κριτηρίων για την ανάθεση της χρηματοδότησης πριν την ένταξη και να διασφαλίσω ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τις χώρες δικαιούχους. Για μένα αυτή είναι μια ε, πολύ σημαντική καινοτομία του νέου μηχανισμού, το οποίο ε, έχει προκύψει από τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις προηγούμενες διαδικασίες διεύρυνσης και θα συμπληρώσει και τα υπόλοιπα μέσα της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω και έναν ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μέσω της ε, χρήσης των κατεξουσιοδότησης πράξεων ε, στη διάρκεια όλης της χρήσης αυτού του μέσου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Βιγγένιν για την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάτσιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ εισηγητά, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ενώπιον μας έχουμε ε, ένα κείμενο που είναι γενικά πολύ καλή πρόταση και βελτίωση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία του προενταξιακού μέσου με το παρόν κείμενο. Και χαίρομαι που ο εισηγητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μη διακρίση, στην προστασία των μειονοτήτων και την καταπολέμηση της δωροδοκίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Συμφωνώ με την επιμονή ε, του ε, εισηγητού για δείκτες ε, απόδοσης. Θα πρέπει αντικειμενικά να μετρούμε για το πώς η βοήθειά μας βοηθάει και τις χώρες αυτές να προοδεύουν στο δρόμο προς την ένταξη. Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, θα ήθελα να σας θυμίσω το τελευταίο δρυμή ψύχος του χειμώνα που οδήγησε σε μεγάλες οικονομικές απώλειες και μέχρι και σε θανάτους ηλικιωμένων. Αυτά τα κρέα φαινόμενα ζητούν ε, άμεση προσαρμογή και είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν μπορούμε πλέον να μιλούμε για συγκράτηση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Αν μπορούν τα δικά μας χρήματα να βοηθήσουν ε, προς αυτή την κατεύθυνση είναι πρόσθετο. Και τέλος θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή να μας διευκρινίσει για ποιο λόγο με τρόπο μάλλον ασυνήθιστο, οι τροπολογίες του για τις κατεξουδιώτηση πράξης ε, υπερβαίνουν τόσα προτείνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σχετικά με αυτό θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο στην ενημέρωση του καταλόγου των δικαιούχων χωρών που δεν ε, είναι αυτό που αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 14 και επαναλαμβάνω ότι δεν ήθιστε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε ένα μέσο ευέλικτο και αποτελεσματικό, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο στη λήψη των αποφάσεων για το ποιο δέχεται προενταξιακή βοήθεια. Ο του Κοινοβουλίου σημαίνει, ε, ε, ε, από την απόφαση σημαίνει και εκτοπισμό των πολιτών και πολιτικά αυτό είναι και εσφαλμένο και απαράδεκτο. Αν μη τι άλλο η Επιτροπή Εξωτερικών θα πρέπει να συμμετέχει άμεσα και δεν μπορεί να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο θα προστίθεται ή θα βγαίνει από τη λίστα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις όχι ο κύριος Ανδρέλης, ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you uh, very much. I will Θα είμαι σύντομος. Καταρχήν, ναι, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βιγγένη. Ε, για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ επίσης και τους άλλους ε, εισηγητές και τους πιο εισηγητές το, των πολιτικών ομάδων και των επιτροπών. Προσπαθήσαμε να μάθουμε, να διδαχθούμε από, το προηγούμενο, από τον προηγούμενο μηχανισμό, να τον κάνουμε πιο απλό, πιο ευέλικτο και αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε σήμερα. Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο εμπλέκεται στην νομοθετική διαδικασία για αυτό το μηχανισμό, αλλά πάντοτε ε, με κάποιο τρόπο συμμετείχε διότι του κοινοποιούνται το, τα έγγραφα στρατηγικής κλπ. Το Δεκέμβριο 2010, αν θυμάστε, είχαμε συνεργαστεί ε, για την διασυνορική συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Οι προτάσει του εισηγητή διευρύνουν τι προτάσει της Κομισιόν, σέβεται παρόλα αυτά το πνεύμα και τη δομή των προτάσεών μας, απλά τις εμπλουτίζει. Κανένα πρόβλημα. Κινούμαστε προ την ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, τονίζει το θέμα της συμμετοχή της κοινωνία των πολιτών, ε, το θέμα της ε, ε, του συντονισμού, της ορατότητας και της παρουσίας στην κοινή γνώμη των δράσεων αυτών κλπ. Ε, το, σε ό,τι αφορά τους στόχους και τους δείκτες είναι επίσης πολύ σωστά τα όσα προτείνει. Το θέμα όμως είναι να ε, μείνουμε ε, ε ευέλικτοι ε, οπότε πρέπει να δούμε τι θα μπει στο στρατηγικό πλαίσιο, τι θα μπει στον κανονισμό και τι θα μπει στα ίδια τα έγγραφα στρατηγικής για να εξασφαλίσουμε αυτή την ευελιξία. Δύο διευκρινήσει. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του μηχανισμού, αναφέρατε αύξηση 23% στον προπολογισμό σε σχέση με το τελευταίο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Σωστό. Με τρέχουσες τιμέ, Ο προπολογισμό που προτείνουμε πάντω είναι ο προπολογισμό του 2013 μείον Κροατία. Και αυτό ο προπολογισμό ε, θα είναι σταθερό για το όλο τον επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει δηλαδή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά είναι σταθερό στα επίπεδα του σταθερός ο προπολογισμό στα επίπεδα του 2013. Αν δείτε τον πληθωρισμό, ε, η πραγματική αύξηση είναι 8% σε σχέση με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι διευκρινιστικά. Για την ε, διασυνορική συνεργασία και το προτινόμενο 7% θα πρέπει να το δούμε. Και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο. Ε, έχουμε ήδη επενδύσει πολλά χρήματα στη διασυνορική συνεργασία, αλλά εδώ η διασυνορική συνεργασία για την οποία μιλάμε είναι ένα τμήμα της ιστορίας, είναι αυτή με τα κράτη-μέλη. Έχουμε και τη διασυνορική συνεργασία μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ε, και της Τουρκίας και αλλού. Προτείνεται μια αύξηση που θα, ε, ε, θα απαιτούσε και από τις έξι δικαιούχες χώρες να επενδύσουν πολύ περισσότερα από εσά, διότι γίνεται συγχρηματοδότηση, άρα έχουν και, αυτά, και αυτές οι χώρες ένα κομμάτι να βάλουν, αλλά θα δημιουργούσε ε, προβλήματα και σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα στην περιοχή. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν αυτή η πρόταση είναι ε, πρακτική και, και ε, βιώσιμη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Κύριος Βικένιν. Πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω τους και για τις παρεμβάσεις τους. Στις επόμενες εβδομάδες πριν την προθεσμία για τις τροπολογίες, θα δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε, διότι πραγματικά επιθυμώ να προτείνουμε ένα κείμενο το οποίο θα υποστηρίζει όλο το Κοινοβούλιο, όλη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μπορούμε να διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα τον εξορθολογισμό των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το αποθεματικό απόδοσης ε, νομίζω ότι ε, λίγο πολύ έχουμε συμπεριλάβει σωστά τι απόψει τη επιτροπή Προπολογισμών για το θέμα αυτό, αλλά μπορούμε να το ξαναδούμε και για τους ε, όρους και τη μερισιμότητα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε λίγο καλύτερα τη διατύπωση, αλλά σε γενικέ γραμμές θεωρώ ότι το θέμα αυτό ε, αντανακλάται καταλήλω στι τροπολογίε που έχουμε προτείνει. Όπω είπα, όμω θα τα ξαναδώ. Όσον αφορά τώρα τα σχόλια του κ. Κάτσι, το βασικό θέμα για τον κατάλογο των χωρών δικαιούχων, αν δεν κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το παράρτημα να είναι κατεξουσιοδότηση πράξη. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο θα έχει λόγο, ε, δεν προτείνουμε αλλαγή, αυτή είναι και η κατάλληλη λύση. Θα μπορούσαμε βέβαια να το ξαναδούμε. Όσον αφορά το θέμα της αλλαγής του κλίματος, εδώ χωράει συζήτηση βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η θέση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου και έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα γιατί ήταν ψυχρός ο περασμένος χειμώνας και δεν μπορώ να, ξέρω, να ξεκινήσω συζήτηση αν όντω υπάρχει αλλαγή του κλίματος προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση, αλλά αν λέμε ότι έχουμε ένα κάποιο ποσοστό των κονδυλίων που σχετίζονται με το μετριασμό των επιπτώσεων του κλίματος, ε, είναι μια σωστή διατύπωση η οποία είναι σύμφωνη και με τις απόψεις ε, των αντίστοιχων επιτροπών. Όσον αφορά τώρα τους δείκτες απόδοσης, ε, μάλλον ξέχασα να σας πω ότι πέραν αυτών των δικτών απόδοσης προτείνουμε η προενταξιακή βοήθεια να περιλαμβάνει και μια αξιολόγηση αντικτύπου στις αιτήσει εκθέσεις πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε να περιλαμβάνεται μια αξιολόγηση αντικτύπου που θα λέει σε ποιο βαθμό και πόσο έχει συνεισφέρει αυτή η προενταξιακή βοήθεια στην πρόοδο των χωρών που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φροντίσω να έρθω σε επαφή και με τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση σήμερα. Ζητώ συγγνώμη ε, και πάλι για τη μικρή μου καθυστέρηση, αλλά ήταν ε, ε, λίγο τρελό το ωράριό μου. Υπήρχε το Κινέζικο Φόρουμ, έπρεπε να πάω και σε μια συνεδρίαση στην Επιτροπή των Περιφερειών και έκανα λάθο υπολογισμό και δεν ήξερα ακριβώ πότε πρέπει να είμαι πίσω εδώ στην αίθουσα. Ελπίζω να με συγχωρέσετε για την καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Ωραία, συγχωρεμένο να είστε στην ώρα σας την επόμενη φορά. Και να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 14η Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Επόμενο σημείο, σύσταση προς το Συμβούλιο για την 67η ε, Σύνοδο της ε, Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εισηγητής ο κύριος ε, Γκραφ Λάμστορφ. Είναι η δεύτερη συζήτηση που γίνεται, δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, για την επέμενη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 36 τροπολογίες κατατέθησαν, συγγνώμη, 136, και ο εισηγητής, ο κύριος Λάμπστροφ, συζήτησε και συμφώνησε με τους κυριώδεις εισηγητές σε 10 συμβιβαστικές τροπολογίες προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο να είναι πιο συνεκτικό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσω και τους κοιόδης ηγητές ε, που εργάστηκαν και τη γραμματεία για το εξαιρετικό του έργο και τις γραμματείες των πολιτικών ομάδων και το προσωπικό. Όπως είπατε ήταν πολλές οι τροπολογίες που κατατέθηκαν και μερικές δικές μου. Ακριβώς γιατί έχουμε περιορισμούς ε, ως προς την έκταση της έκθεσης δεν είχε καλυφθεί η διάσκεψη του Ρίου και η διεθνής δικαιοσύνη και κάτι άλλα επίκαιρα θέματα. Επίσης είναι σημαντικό ότι λάβαμε γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης, ε, ΔΕΒΕ, και μπορούμε να πούμε ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Ε, ουσιαστικά και μεγάλα τμήματα της γνωμοδότησης τους θα τα εντάξουμε και στη δική μας έκθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες αφορούν κυρίως ζητήματα ευρεία αποδοχή και συνένεση. Ευθύνη για προστασία, διεθνή δικαιοσύνη, γυναίκε σε μόλεμε σειράξει κτλ. Αλλά και περιβαλλοντικά ζητήματα που συμπεριλαμβάνει και τη διάσκεψη του Ρίου και κάτι άλλο που είναι σημαντικό για του συναδέλφου και εδώ και τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Ε, η διαδικασία μετά το 2015 ε, και οι στόχοι ε, της ε, χιλιετίας και η διαδικασία αυτή. Η μία αναπτυξιακή στόχη για το πώς θα είναι στόχοι που θα έχουν οριστεί με καλό τρόπο και θα μπορούν να ανακοινώνονται. Υπάρχει μια πρόταση της Βραζιλίας να γίνει συζήτηση για την ευθύνη κατά τη διάρκεια της προστασίας. Κανείς δεν γνωρίζει ε, ποια κατεύθυνση θα πάρει τελικά αυτή η συζήτηση, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η ευθύνη για προστασία είναι ένα δόγμα που αναπτύχθηκε το 2005 και θεωρούμε χρήσιμο και στο διεθνές δίκαιο και για τη μεταξέλιξη του διεθνούς δικαίου. Εδώ είμαστε λίγο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Ένα θέμα που επανέρχεται και είναι επίμαχο είναι ο ρόλος των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων ε, στις εργασίες των ΗΕ. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι ε, στο οποίο έχουμε ε, μια τροπολογία. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί, όπως γνωρίζετε όλοι. Και ήδη Έχω στείλει κατάλογο ψηφοφορία με τις ενδείξεις μου. Ε, ελπίζω ο πρόεδρος να με ακολουθήσει. Αν έχετε αφιβολίε, ερωτήσεις για οποιαδήποτε ειδική τροπολογία. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και πάλι και προσβλέπω στην ψηφοφορία. Ήταν υποδειγματική συνεργασία. Ευχαριστώ. Σκιώδης τώρα. Κορίνα Κρέτου. Κυρία Κρέτσου, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ τον κύριο Λάμστορφ και τους συναδέλφους μου της ομάδας των Σοσιαλιστών, ιδιαίτερα της, και την κυρία Μουνής και τον κύριο Λάινεν. Η συζήτηση λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο ε, των λειτουργικών αδυναμιών του, ΟΕΕ που γίνονται όλο και πιο προφανείς και ορατές. Για παράδειγμα, στη Συρία λαμβάνει η χώρα ε, σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και οι συστήσεις που γίνονται στην, ε, στον Εθνών δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να προωθήσουν δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, αυτό είναι η υποχρέωσή μας πλέον. Η θέση μας έχει ως στόχο να βελτιώσει την συνεκτικότητα ε, της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ορατότητά της. Θέλουμε να είμαστε ένας ορατός παίκτη στο επίπεδο των ΗΠΑ χρειάζεται μόνο ένα ευρωπαϊκό μήνυμα να περνάει με εναρμονισμένη θέση όλων των κρατών μελών. Ε, τονίζουμε επίσης την σημασία βελτιωμένου συντονισμού, της ε, διαφάνειας και της ανταλλαγής ε, πληροφοριών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δύο συστάσεις αφορούν την βελτιστοποίηση της, ε, του αντικτύπου της δράσης μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και α, η αρχή είναι αποτελεσματική, αποτελεσματική πολυμέρεια. Νομίζω ότι έτσι θα νομιμοποιηθεί η ε, θέση μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να βελτιωθεί, για να επιτευχθεί αυτή ε, η νομιμοποίηση θα πρέπει να νομιμοποιηθεί περισσότερο και ο ΙΕ με μεταρρύθμιση του. Ε, θα πρέπει να δοθεί μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Συμβούλου Ασφαλεία και να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΗΕ για να βελτιωθεί η δημοκρατική φύση, η διαφάνεια και η αξιοπιστία του Παγκόσμιου Μηχανισμού Διακυβέρνησης. Ευχαριστώ τον κύριο Λάμστορφ γιατί συμπεριέλαβε και το θέμα της ανάπτυξης στην έκθεσή του. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ο πιο σημαντικός δωρητής ε, ε, ε, ε, συγγνώμη, πιο σημαντικός ε, συνεισφορέας στον προπολογισμό του, του ΟΗΕ, είναι περίπου στο 30% του συνολικού προπολογισμού, οπότε ε, έχουμε πιο σοβαρό λόγο. Any other ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις? Κύριε Λάπτο. Με ναι, μπορώ παρά να ευχαριστήσω και την Κορίνα και τους άλλους συναδέλφους. Πιστεύω ότι αύριο η ψηφοφορία θα βοηθήσει και τους συναδέλφους να καταλάβουν το εξής. Με την αυριανή ψηφοφορία θεωρούνται οι συστάσεις εγκεκριμένε, εκτό αν μια άλλη πολιτική ομάδα τα θέσει νέες πράγμα που δεν αναμένω γιατί δεν εκφράστηκε τέτοια επιθυμία στο παρελθόν, ούτε ξαναγίνει. Και χρονικά είμαστε εντάξει. Το Συμβούλιο θα συζητήσει αυτά τα θέματα σε ένα μήνα και αν αύριο το εγκρίνουμε, θα το παρουσιάσω στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τα Ηνωμένα Έθνη για περαιτέρω εξέταση. Και είναι μια πολύ καλή διοργανική συνεργασία. Σα ευχαριστώ. Και τώρα τι κάνουμε. Θέλετε το λόγο κύριε Πρέντα. Γιατί είχαμε ολοκληρώσει τη συζήτηση. Εν πάση αν θέλετε το λόγο. Σας είπα ότι αυτή η, σύνοψη δεν ήταν ολοκλήρωση συζήτηση, ήταν διάμεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο να πω και εγώ μερικά πράγματα. Συνεργάστηκα θαυμάσια με τον κύριο Λάμστορφ. Ελπίζω να συμφωνεί και ο ίδιος με τα λεγόμενά μου. Κοιτάζω τον κατάλογο ψηφοφορίας που μας έστειλε χτες το απόγευμα. Βλέπω ότι ο κύριος Λάμστορφ Διαφωνεί με πολλές από τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η πολιτική μου ομάδα. Το καταλαβαίνω προφανώς ότι έχει διαφορετική προσέγγιση. Αλλά Εγώ με τη σειρά μου υποστηρίζω τις περισσότερες προτάσεις του εισηγητού και ε, τις περισσότερες υποδείξεις για τις τροπολογίες, αλλά δυστυχώς ούτε εγώ ούτε η ομάδα μου ε, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ε, τροπολογίες 8 και 10. Αυτές οι τροπολογίες συμβαστικές αφορούν ε, τροπολογίες που είχαν καταθέσει μέλη άλλων πολιτικών ομάδων και κανένα μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν είναι διατεθειμένο να υποστηρίξει τις συμβιβαστικές 8 και 10. Επίσης, το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας 8 δεν αντιστοιχεί με την ε, θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα όταν εγκρίναμε το ψήφισμα για την οδηγία του Συμβουλίου για ένα κοινό σύστημα ε, φόρων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και εδώ σκέφτομαι ιδιαίτερα την αιτιολογική σκέψη α. Οι τροπολογίες 136 και 135 αφορούν τη δημιουργία κοινοβουλευτικής συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και επειδή ούτε ο εισηγητής ούτε οι σκιώδεις εισηγητές ε, δέχτηκαν αυτές τις τροπολογίες, εμείς προτείναμε μια συμβιβαστική λύση, δηλαδή να εγκριθεί προφορική τροπολογία για τη σύσταση κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δυστυχώς ε, ούτε σε αυτό συμφώνησαν όλοι οι συντάκτε των τροπολογιών. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι εμεί θα καταψηφίσουμε τι τροπολογίε 135 και 136. Ζήτησα επίσης δύο τροπολογίες κατά τμήματα, ε, η 128 τροπολογία που είναι του εισηγητού και μία ε, άλλη ζητούμε να ψηφιστούν ξεχωριστά. Ευχαριστώ και πάλι κύριε ε, Λάμστορφ. Ο κύριος Λάινεν. Yeah, Ο έχασε τώρα το μάτς, το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή την έκθεση την κερδίζει κάθε χρόνο. Θα επανέλθω όμως στη δική μου τροπολογία που είχα κάνει μαζί με άλλους και πέρσι και φέτος υπέρ του εκδημοκρατισμού των Ηνωμένων Εθνών με μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινοβουλίων εν γέννη. Το θέμα θα επανέρχεται ξανά και ξανά γιατί είναι πάγιο. Αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι πέρσι είχαμε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της κοινοβουλευτικής συνέλευσης με παγκόσμιο απόϊχο. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 15 μέρες ήμουν στο Νέο Δελχή ε, και 50 βουλευτές ε, της Ινδικής Βουλής ε, ζήτησαν τα ίδια. Και στη Σενεγάλη επίσης και ο νέος Πρόεδρος και το Κοινοβούλιο είναι υπέρ αυτής της άποψης. Θα ήταν μεγάλη αποδυνάμωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν οι τροπολογίες αυτές 135-136 απορριφθούν. Και τι έχει αλλάξει από πέρσι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Για αυτή τη μεταστροφή η δική μου πολιτική ομάδα θα τις υπερψηφίσει. Επίζω η πράσινη, η φιλελεύθερη δεν ξέρω. Κατά τα άλλα συμφωνώ σε όλα με τον Αλεξάνδρ Λάμστροφ αλλά είναι διπλωμάτης και ξέρω ότι οι διπλωμάτε και το καταλαβαίνω δεν αγαπούν τα κοινοβούλια και το είπα και συζήτησα και με διπλωμάτε και με το δικό μου πρέσβη και λέει αυτό μας έλειπε τρόμος να προσθεθεί και κοινοβούλιο τώρα στον ΟΗΕ. Αλλά θα πρέπει οι πολίτες να έχουν στην παγκόσμια πολιτική φωνή και θα έρθει κάποια στιγμή αυτή η ώρα. Και η IPU, η Διεθνής Κοινοβουλευτική Ένωση, δεν είναι υποκατάστατο είναι ένα σύνολο, ένα, μια συνέλευση των κοινοβουλίων επί παντών επιστητού. Ούτε είναι όργανο του ΟΗΕ, ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ. Έχει καθεστώς παρατηρητή σαν την Greenpeace. Μα είναι γελίο τα κοινοβούλια να είναι παρατηρητές, δηλαδή στον ΟΗΕ, θεατές και καμιά φορά να παίρνουν και το λόγο άμα τους το δίνουμε. Αυτό είναι, αυτά είναι τελείως γελία πράγματα. Και παγκοσμίω συμμετέχω και εγώ σε αυτή την εκστατεία με άλλους πολλούς στο κοινοβούλιο. Η μεγάλη υποστήριξη... Ε, κοινοβούλιο, αφρικανικό, ε, λατινοαμερικανικό και τώρα το Ινδικό. Αν αύριο πάει στραβά η ψηφοφορία, θα φανούμε τελείως αναντίστοιχοι, ε, αναξιόπιστοι και αναντίστοιχοι. Δεν ξέρω τι διατύπωση. Αλλά τι θα πούμε, φέτος, ξέρετε, αλλάξαμε γνώμη και είμαστε κατά. Ενώ πέρσι ήμασταν υπέρ. Είναι τελείως γελία αυτά τα πράγματα και βλακίες και δεν ξέρω ποιος τα ανακοινεί και τα ανακατεύει. Καινούργοι ε, που δεν έχουν καμία ιδέα για το τι συνέβη πέρσι και ε, απορρίπτουν, αποσύρουν περσινές αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος με όλα αυτά. Ευχαριστώ. Last. Στη συνέχεια, τελευταίος ομιλητή, τελευταία ομιλήτρια η κυρία Λοκπίλερ από τους Πρασίνους. Ε, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Η Φρανσίσκα Μπραντνερ είναι η σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα μας, αλλά νομίζω ότι μπορώ να πω και από πλευρά τη ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε καταλήξει στη συμβαστική πρόταση 3, διότι καθορίζει τον την εφαρμογή του ρόλου των γυναικών ε, ε, στην ε, ειρήνη και την ασφάλεια. Έχουν συμπεριληφθεί πολλά από τα όσα έχουμε προτείνει γενικώ στο κείμενο και από τις υπόλοιπες τροπολογίες που καταθέσαμε Νομίζω ότι πολύ συχνά περιγράφεται τι εννοούμε σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα συνεχίσουμε να τι καταθέτουμε. Και σας ευχαριστώ για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριο Λάμπστροφ. Ναι. Καταρχάς να πω ότι εμένα μου αρέσει το κοινοβούλιο. Ήμουν διπλωμάτης. Σήμερα είμαι ποδοσφαιριστής. Έχασα από την Πορτογαλία. Σας είδαμε να παίζετε, λέει ο κύριο Προβερά, αλλά κερδίζω ε, στην έκθεση, οπότε κάτι πήρα κι εγώ σήμερα. Καταρχάς, λοιπόν, να σας πω για τι συμβαστικέ προτάσεις 8 και 10, το ΕΛΚ μας ενημέρωσε εκ των προτέρων ότι δεν θεωρούν ότι εκπροσωπούνται καταλήλως ε, σε αυτή τη συμβαστική πρόταση και θα την καταψηφίσουν. Το ελέγξαμε με τους άλλους ε, σκιώδεις συζητητές. Ε, τους υποστηρίζουμε και θα δούμε κυρίως τα θέματα της περιβαλλοντικής ε, διακυβέρνησης. Για την 122 θα πρέπει να τη δω, δεν θυμάμαι ποια ήτανε. Ε, νομίζω ότι θα ψηφιστεί όμως. Τώρα, για το θέμα αυτό το διαβόητο της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, για μας είναι σημαντικό το θέμα, γιατί δεν είναι επανομοιότυπα τα δύο στοιχεία. το Κοινοβούλιο έχει την ελευθερία να αποφασίζει για τα θέματα αυτά, διότι όπως είπε και κάποτε ο Κόρνετ Αντενάουερ, ακόμα και οι πολιτικοί μου αντίπαλοι δεν μπορούν να με αποτρέψουν από το να γίνομαι πιο ευφυής κάθε μέρα. Εάν φέτος λοιπόν έχουμε μια ψηφοφορία με διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτό θα δείξει ότι είναι ζωντανή η συζήτηση και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πάντα γίνεται ιδιαίτερα ζωντανή συζήτηση. Ε, η περισσότεροι συμφωνούμε στο 99% των θεμάτων που αφορούν τον ΟΗΕ, διαφωνούμε στο 1%. Εάν δημιουργηθεί η κοινοβουλευτική συνέλευση θα δούμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Καταρχάς θα πρέπει να εντοθεί στον ιδρυτικό χάρτη και στο σημείο 2 δηλαδή τη ισότητα των κρατών μελών των Ηνωμένων Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα θα μπορεί να ορίσει αυτό που θεωρεί κοινοβούλιο για να συμμετέχει σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση. Ε, θα συμμετέχει για παράδειγμα το Κογκρέσο των Κινέζων, ε, το, οι Βορειοκορεάτες επίσης θα εκπροσωπούνται και ούτω καθεξής. μία μειοψηφία κοινοβουλίων παγκοσμίω έχει εκλεγεί δημοκρατικά με τον τρόπο που το εννοούμε εμεί. Επομένως, αυτή η κοινοβουλευτική συνέλευση δεν μας, θα μας οδηγήσει αυτόματα στον εκδημοκρατισμό των Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι όπω σα είπα στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά μόνο στα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ε, τα κυρίαρχα κράτη και τα κοινοβούλια τους. Υπό τη λογική λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών, εμείς δεν είμαστε ένα κυρίαρχο κοινοβούλιο, διότι δεν είμαστε κοινοβούλιο ενός κράτους και επομένως δεν είμαστε μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα ήμασταν εκτός αυτής της διαδικασίας και θα βρισκόμασταν να χτυπάμε στην πόρτα της συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνέλευσης και να ζητάμε καθεστώς παρατηρητή, κάτι το οποίο στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα περιγράφει ως γελίο τουλάχιστον. Νομίζω λοιπόν ότι από δημοκρατική σκοπιά ε, σε γενικές γραμμές, αλλά και από θεσμική ε, άποψη, ε, ε, εσωτερική εδώ του κοινοβουλίου μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να πιέζουμε αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να συνεργαστούμε. Έχουμε αιτήσει αντιπροσωπεία στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μας συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά οι εταίροι μας και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε επίπεδο πρεσβειών κατών μελών και έχουμε και πολλά να αποκομίσουμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορούμε να προβλέψουμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση. Οι εθνικέ αντιπροσωπείς που πηγαίνουν στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνουν και βουλευτέ. Κανένα κράτο μέλο δεν απαγορεύεται να το κάνει. Μπορεί κάλλιστα κάποιο να στείλει βουλευτέ και μπορεί και αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου ή και φέτο να συμπεριλάβει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αντιπροσωπεία τη ακριβώ για να ενισχύσουν το ρόλο τη. Υπάρχουν λοιπόν πάμπολοι τρόποι να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική πτυχή των εργασιών των Ηνωμένων Εθνών χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου δεν είναι και το πλέον δημοκρατικό ε, όργανο και είναι και μάλλον δαπανηρό. Συνεπώς θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικού τρόπους με τους οποίους είχαμε και επιτυχία στο παρελθόν και έχω και την άποψη ότι μακροπρόθεσμα η ενίσχυση της Διεθνής Κοινοβουλευτικής Ένωσης ε, θα είναι κάτι καλύτερο διότι ε, ε, υπάρχουν κάποια θέματα νομικής φύσεως ορισμένες φορές θεωρούνται υποδεώστερα τα κοινοβούλια από τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής θα πρέπει λοιπόν να βρούμε εναλλακτικού τρόπους και όχι να δημιουργήσουμε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση των ΗΠΑ βεβαίως δεν θα πρέπει να είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας τέλος να σας πω ότι εμένα μου αρέσουν τα κοινοβούλια μου αρέσουν τα όσα κάνουμε εδώ, όπως διαπιστώνετε. Πολλές φορές κατορθώνουμε να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα. Κάποιες φορές υπάρχουν διαφωνίε, αλλά είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίε και μάλιστα γίνονται και σε λογικά πλαίσια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε τις 135 και 136 και θα δούμε ποιος θα κερδίσει αύριο στην ψηφοφορία. Ε, σήμερα μας κέρδισε η Πορτογαλία, μπορεί αύριο να κερδίσω εγώ. Thank you. Ευχαριστώ. Συμφωνώ 100% μαζί σας. Συμπορία πήρε. Mm, yes, okay. Yeah. Just a few words because... Δυο λόγια μόνο, γιατί μην ξαναξυχήσουμε τη συζήτηση. Λάμστορφ lost 4-2 in football. Έχασε 4-2 ο Λάμστορφ στο ποδόσφαιρο. Now he has to win 5-1. Uh, Τώρα θα πρέπει στον επαναληπτικό να κερδίσει 5-1, γιατί αλλιώ δεν θα, μας, δεν θα ισοφαρίσει. I'm really astonished. Με εκπλήσουν τα επιχειρηματά σου, Αλεξάνδρ. Μια αντιπροσωπεία του ΕΛΚ ε, πήγε στη Νέα Υόρκη και έχω πάει μαζί σου στη Νέα Υόρκη και αυτό το χρησιμοποιείται το χρησιμοποιείς ως επιχείρημα εναντίον της ε, κοινοβουλευτικού, οργάνου ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας που παρακολουθεί στενά όλα, όλες τις εξελίξεις. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. η Κοινοβουλευτική Ένωση έχει άλλη φύση. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει τμήμα του ΟΗΕ. Η Κοινοβουλευτική Ένωση έχει ο, έδρα τη Γενέβη και μετακινείται για τρεις μέρες το χρόνο στην, στη Νέα Υόρκη. Ε, δεν πρόκειται για όργανο του, ε, του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Θα, μπορούσα, θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιηθεί το άρθρο 22 και με πλειοψηφία να ε, δημιουργηθεί αυτό το όργανο. Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Θα έπρεπε να μείνει ανοιχτή αυτή η πόρτα της μεταρρύθμισης ε, πλέον στην παγκοσμιοποίηση, στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ε, θα πρέπει να φτάσουμε στους πολίτες, όχι μόνο στους διπλωμάτες και τους πολιτικούς. Ε, ε, αν διαφωνήσουμε με τη δημιουργία της κοινωνιστικής συνελευσής είναι σαν να αρνούμαστε στους πολίτες συμμετοχή. Ξέρω ότι οι διπλωμάτες δεν αρέσκονται, δεν, μάλλον στους διπλωμάτες δεν αρέσουν τα κοινοβούλια, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Να απαντήσω εν συντομία. Δεν αναφέρθηκα μόνο στην αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ. Η Ντροά επίσης πηγαίνει στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι συνάλφοι Τη Επιτροπή ανάπτυξη επίσης μιλούν στην, στο πρόγραμμα, πρόγραμμα του ΟΗΕ, του UNDP κλπ. Ακόμα και η Επιτροπή ε, ε Δημοσιονομικού Ελέγχου πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να συζητήσει με του ελεγκτές. Συνεπώ πολλά πράγματα συμβαίνουν. Και τέλο. Ε, ε, η ε, σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση έτσι κι αλλιώς οι εκπρόσωποι θα ήταν εθνικοί εκπρόσωποι. Ε, συνεπώς ακόμα και μια τέτοιου είδους κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού δεν θα μπορούσε πράγματι να ελέγξει ε, τις, ε, ε, τις χώρες τις ίδιες που συμμετέχουν. We'll at... Σας ευχαριστώ. Αύριο η ψηφοφορία είναι στις 12 ε, παρατέταρτο. Και τώρα ακολουθεί διάλειμμα μέχρι τις 5.30.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ε, της Μολδαβίας, τον κύριο Λεάνκα, για ανταλλαγή απόψεων. Καλωσορίζουμε και κυρία Μακοβέη, πρόεδρο της ε, Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Να ξεκινήσουμε αμέσως ε, τη συνάντηση αυτή και να σας πω ότι είχε ευτυχές ε, ξεκίνημα η φετινή χρονιά. Ο πρόεδρος Τιμόφκη εξελέγει στις 16 Μαρτίου ε, και με αυτό έληξε η συνταγματική κρίση η οποία είχε διάρκεια δύο ετών. Υπήρξε μια μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας και ξεκίνησαν και οι διαπραγματεύσεις για θέματα εμπορίου, ε, κυρίως για θέμα ελευθέρωση συναλλαγών και Υπάρχει μια μακρά συνεργασία. Ο διάλογος για τις θεωρήσεις διαβατηρίων είναι σε καλό επίπεδο και η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετική. Τέλος, οι διαπραγματεύσεις με τη Σπολ ε, συνεχίζονται σε άτυπο επίπεδο. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Μαΐου επισημαίνει ότι έχει γίνει καλή πρόοδο σε όλα τα σημεία του προγράμματος δράσης, αλλά σημειώνει κάποιες καθυστερήσεις στην έγκριση σημαντικού τμήματος νομοθεσίας και ε, πολλά θέματα εφαρμογής και υλοποίησης των όσων προβλέπονται στην νομοθεσία αυτή. Στην έκθεση τη καλεί τη Μολδαβία να κάνει περαιτέρω προσπάθεια ε, για τα θέματα τη δικαιοσύνη και τη μεταρρύθμιση ε, στον τομέα της δικαιοσύνης, να συνεχίσει το διάλογο για να καθορίσει μηχανισμούς για την εφαρμογή των ε, δραστηριοτήτων δημιουργίας εμπιστοσύνης και να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες έγινε η τρίτη συνεδρίαση στα πλαίσια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας και ένα από τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν ιδιαίτερα ήταν η νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Θα σταθώ σε αυτό εγώ. Σας δίνω ε, χρόνο λοιπόν ομιλίας, αγόρευσης και θα ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτά που έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω ε, την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δίδεται να μιλήσω ενώπιον ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στη Μολδαβία και την περιφέρεια, της προκλήσης που αντιμετωπίζουμε, καθώς επίσης και τις προοπτικές. των σχέσεων Μολδαβίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που βλέπουμε εδώ και τον πρόεδρο Μπούζεκ, και πάλι εξ ονόματος της κυβέρνησής μας θα ήθελα να εκφράσουμε τη βαθιά μας ε, ευγνωμοσύνη για το ε, σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε για ε, να φτάσουμε εδώ και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας, μας βοήθησε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μακοβέη για το καταπληκτικό της έργο ως πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, αισθανόμαστε ότι μας υποστηρίζει και μας ε, καθοδηγεί και είμαι αισιόδοξο όταν βλέπω τόσο ενδιαφέρον και τόση υποστήριξη από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, και πρέπει να σας πω ότι ερχόμενος εδώ δεν είναι πρώτη φορά που έρχομαι Είχα ξανάρθει πριν από τρία χρόνια, το Μάιο του 2009. Έγιναν εκλογές τον Απρίλιο και ε, συμπίπτει αυτή η τριετία ε, από την ανάλυση περίπου των καθηκόντων των κυβερνητικών του συνασπισμού που είναι ο συνασπισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να σας πω ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι και οι προτεραιότητες ε, της ε, κυβέρνησης. Πολύ σύντομα να θυμίσω που βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Ήταν μια χώρα με ε, ένα αυταρχικό καθεστώς ολοκληρωτικό, μια χώρα που είχε πάρει ένα κατήφορο προς τους θεσμούς της. Η διοίκηση χρησιμοποιεί το για να πολεμήσει την αντιπολίτευση και όχι μόνο για να παραβιάσει τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα για καταστολή. Ε, ήταν σε σχέση κρίσης με τους δύο γείτονες, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Η χώρα βρισκόταν σε μια κατάσταση αναστολής των σχέσεων με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είχε αποφασίσει η κυβέρνηση να επιβάλλει θεώρηση διαβατηρίων στους Ρωμάνους πολίτες, δηλαδή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε κάποιο βαθμό η χώρα αυτό απομονωνόταν και σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που αποχώρησε ε, τον Ιούνιο του 2009 χωρίς να είναι σε θέση να βοηθήσει ε, και την οικονομική κατάσταση. Ε, η ύφεση τότε ήταν 7% και μείον 16% το έλλειμμα του προπολογισμού σχέση με το ΑΕΠ. Τρία χρόνια μετά αυτές τις δραματικές αλλαγές ε, στην ηγεσία της χώρας έρχομαι να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ε, ένας συνάδελφος από το Ίδρυμα Ανοιχτή Κοινωνίας μου έδωσε αυτό το έγγραφο που είναι πάρα πολύ σημαντικός δείκτης για το πού βρίσκεται σήμερα η Μολδαβία είναι ένας ε, κατάλογος ε, της ευρωπαϊκής προοπτικής ε, των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών που είναι μέλη της Ανατολικής Γειτονίας δηλαδή. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστο αυτό το έγγραφο για το πώς προχωράει η οικοδόμηση της δημοκρατικής κοινωνίας στις χώρες αυτές και πώς μπαίνουν τα θεμέλια μιας ελεύθερης και σταθερής κοινωνίας και με χαρά μαθαίνω ότι πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια η Μολδαβία. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι το 2009 σε κάποιο ε, βαθμό η Μολδαβία ήταν ο απόκληρος της ανατολικής ε, γειτονίας. Είχε πάρα πολύ κακές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες σχεδόν ε, και στις παραμέτρους ελευθεροτυπία, ας πούμε, αντιμετώπιση του κράτους ε, ως προς τα ε, βασικά θεμελιώδη δικαιώματα και σε αυτή την τριετία κατάφεραν να ε, επιτελέσει τεράστια πρόοδο η κυβέρνηση της Μολαβίας. Μεγάλη αλλαγή επήλθε στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα πολιτικά όργανα και οι θεσμοί, η οικονομία και επίσης έχει έρθει και μεγάλη αλλαγή στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποια πρόοδο, αυτό οφείλεται στις πολύ καλές σχέσεις και στην ε, πρωτοφανή προθυμία με ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Κάναμε βέβαια κάποια πρόοδο, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τεράστιες ε, προκλήσεις. Βεβαίως, πριν από δύο μήνες εκλέξαμε πρόεδρο και δεν είχαμε πρόεδρο για 917 ημέρες. Και ε, άρχισαν ε, διάφορες φιλοσοφικές συζητήσεις σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Μήπως είναι ε, ξεπερασμένος ο θεσμός της Προεδρίας. Χρειαζόμαστε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βεβαίως αστείευομαι. Τώρα ε, υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο και έχουμε ακόμα μια τριετία μέχρι τις επόμενες εκλογές και μπορεί η κυβέρνηση να επικεντρωθεί σε πάρα πολύ δύσκολες όσο και απαραίτητες όμως μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζετε ποιες είναι οι ευαίσθητες μεταρρυθμίσεις και οι τομείς ε, κλειδιά για την κυβέρνηση. Ε, αναθεώρηση και μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ε, των αρχών επιβολής του νόμου, ε, της οικονομίας και εδραίωση των θεσμών. Είναι βασικοί οι τομείς και προτεραιότητε και συνδέονται πάρα πολύ με τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε, η δικαστική μεταρρύθμιση, η αστυνομική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση της εισαγγελία, όλοι αυτοί οι στόχοι συνδέονται ε, με ε, το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ε, θεωρήσεις διαβατηρίων. όλα αυτά τα θέματα, καταπολέμηση της διαφθοράς, τα θέματα των επίκορων. Χαίρομαι ε, που βρίσκομαι στις Βρυξέλλες ε, ε, μετά την ολοκλήρωση της νομικής προσέγγισης. Κρίναμε 42 νόμους και αποφάσεις στη κυβέρνηση σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης για τη θεώρηση διαβατηρίων. Ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν οι αντιστάσεις ορισμένων κλάδων της κοινωνίας και θεσμών. Πάντως ε, η κυβέρνηση έδειξε αποφασιστικότητα να πολεμήσει ορισμένες προκαταλήψεις που ισχύουν στην κοινωνία για να ε, ε, οικοδομήσει μια κοινωνία πιο ανεκτική, πιο ευρωπαϊκή που να βασίζεται στις κοινέ μας αξίες. Είπα ότι οι προκλήσεις παραμένουν και στην οικονομική ανάπτυξη. Δυστυχώς η Μολδαβία σύμφωνα με τις στατιστικές είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη παρόλο που το 2010 και το 2011 ε, το έλλειμμα του προπολογισμού ήταν 6,4%, ε, φτάσαμε στο 2,4% ε, και το σημαντικότερο είναι ότι ο πρώτος εμπορικός εταίρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 52% του εξωτερικού μας εμπορίου πηγαίνει προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ ε, μεγάλη η ε, πρόοδος ε, της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μειωθεί η ανάπτυξη σε 3%. Ξέρω ότι στις χώρες σας 3% είναι πολύ ωραίος ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας. Εμείς δεν μπορούμε όμως να το θεωρήσουμε επιτυχία γιατί έχουμε αρχίσει από πολύ χαμηλότερο επίπεδο να αναπτυσσόμαστε. Ε, ξέρετε ότι υπάρχει το θέμα της ε, διένεξης της υπερβνηστερίας. Ε, πρέπει να σας ενημερώσω ότι είναι θετικές οι προοπτικές μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε πολύ επικοδομητικό διάλογο για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο όχθεων του Δνύστερου δημιουργούμε ένα περιβάλλον που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη λύση. Ε, υπάρχει και η προθυμία για οικονομική ενίσχυση. Ξέρουμε ότι ε, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να λυθεί αυτή η διένεξη. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω πάρα πολύ στην εισαγωγή μου. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν έχουμε ευρωπαϊκή προοπτική, δεν είναι ακόμα επιλέξιμη για τη διεύρυνση της Ένωσης. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψήφισμα που εγκρίνατε πέρσι το Σεπτέμβριο. Ήταν το πρώτο έγγραφο που είχε τέτοιο σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τονίζει και παραπέμπει στο άρθρο 49 της συνθήκης που αναγνωρίζει της Λισαβόνας δηλαδή, ότι οποιαδήποτε χώρα που ε, τηρεί κάποιες προδιαγραφές και είναι ευρωπαϊκή έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ε, για ένταξη και ήταν πολύ ισχυρή ενθάρρυνση και ηθική ανάταση μας έδωσε. Ε, υπάρχει δυνατότητα πλέον ε, να είναι υποψήφια χώρα η Μολδαβία για διεύρυνση και θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό, αν έχουμε την ευκαιρία ή όχι. Και το έγγραφο που σας δείχνω αναγνωρίζει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο και η Μολδαβία είναι πλέον ο καλός μαθητής στην Ευρώπη. Και μαζί μπορούμε να σας δείξουμε ότι μπορούμε ε, στη γειτονιά μας που είναι πάρα πολύ δυναμική και αναπτυσσόμενη ε, να βοηθήσουμε. Δεν είναι πάντα θετικός αυτός ο δυναμισμός. Σήμερα υπογράψαμε με την Επίτροπο Γεωργίευα ε, ειδικέ διατάξεις για την πρόληψη των θεομηνιών και πολύ συχνά στη δική μας περιοχή ε, δεν είναι θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές, είναι ανθρωπογενείς. Μόνοι μας τις ε, προκαλούμε. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι να μην φαινόμαστε απλώς Ευρωπαίοι, αλλά φερόμαστε και ως Ευρωπαίοι και να αντιδρούμε ως Ευρωπαίοι. και παρακαλώ να αναγνωριστεί και η ευρωπαϊκή προοπτική μας γιατί έτσι θα μας δοθεί ένα κίνητρο, μια ενθάρρυνση να, να εμπιστευόμαστε περισσότερο τις δυνάμεις μας και πάλι με τη δική σας γενναιόδορη υποστήριξη θα διευρυνθεί η σταθερότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο προς Ανατολάς. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως προσβλέπω ε, στις ερωτήσεις να απαντήσω με χαρά. Ευχαριστώ yeah, Ευχαριστώ πολύ για αυτή, αυτή την ε, γεμάτη πάθος ε, ε, παρουσίαση. Ο πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας, ο κύριος ε, Μακο... η κυρία Μακοβάη, συγγνώμη. ορίζω τον Υπουργό. Ε, συνεργαζόμαστε εδώ και δυόμιση χρόνια μαζί του. Χτες σας ενημερώνω ότι έλαβε χώρα η συνεδρία Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και υιοθετήσαμε και κάποιες συστάσεις τις οποίες θα, των οποίων θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή. Θα ξανασυναντηθούμε στο Τσισινιό τον Οκτώβριο. Ε, τρία βασικά θέματα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μολδαβίας, ε, η Συμφωνία Σύνδεσης, οι θεωρήσεις ε, και και η Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορίου. Ε, οι ε, συνάδελφοι από την Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων που εργάζονται για αυτό το θέμα έχουν αναφέρει πολύ καλή πρόοδο ε, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης. Ε, μόνο ένα κεφάλαιο είναι ανοιχτό, μόνο το περιβάλλον, το οποίο θα κλείσει και αυτό σύντομα από ό,τι φαίνεται. Επίσης και σε ό,τι αφορά τις, ε, τα άλλα δύο θέματα της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και της, ε, των θεωρήσεων έχουμε θετικά μηνύματα. Πριν από... Ε, μπορούμε να, να αναλογιστούμε ποια ήταν η κατάσταση πριν από τρία χρόνια και ποια είναι τώρα. Οι τεχνικοί που παρακολουθούν τι διαπραγματεύσει μα λένε ότι πολλέ φορέ η Μολδαβία κινείται τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Ε, Προφανώ θα πρέπει να επιβραβευθεί. Ε, πάντοτε η αρχή που ακολουθούμε είναι περισσότερα για περισσότερα. Σίγουρα δεν θα πρέπει να παίρνουμε όλες τις χώρες μαζί ε, σαν να είναι μια δέσμη. Θα πρέπει κάθε χώρα να επιβραβεύεται ανάλογα με τις επιτυχίες της. Αυτό που συμβαίνει άλλωστε στην καθημερινή μας ζωή. Σίγουρα απομένει πολύ έργο μπροστά μας, μπροστά σας. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε όπως και τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, ακόμα και ιδιαίτερος με κλεγμένο πρόεδρο πλέον. Ε, μία σύσταση που περιλαμβανόταν και στην περσινή έκθεση είναι η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την υπερνηστερία, αντικατάσταση με ε, πολιτοφυλακή διεθνή, πολιτοφυλακή ε, Επίσης θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα πυρομαχικά και ε, τα οπλικά συστήματα που υπάρχουν και ε, επίσης ε, χτες αναφερθήκαμε στο θέμα της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφοριών έτσι ώστε να έρθουν στα ευρωπαϊκά επίπεδα να λειτουργούν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτά. Στη συνέχεια, ο κύριος Γκραμ Βότσον δεν είναι εδώ. Ο κύριος Πρόεδρος, κύριε Μπούζεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, κύριε Αναπλήρωτη Πρωθυπουργέ, για όλα όσα έχετε καταφέρει στη χώρα σας ε, το τελευταίο διάστημα αποτελεί τη χώρα πρότυπο. Στο ανατολικό τμήμα της Υπήρους μας, από τη δική μας οπτική γωνία. Δεν θα θέλαμε να σας πιέσουμε βεβαίως να κάνετε τίποτα, γιατί τα πάντα πρέπει να είναι δική σας απόφαση. Αν αλλάξει το οτιδήποτε στη χώρα σας, θα πρέπει να τα αποφασίσετε εσείς. Αυτό όμως προσδοκούμε. Η απόφαση όμως επαφείται σε εσάς. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μια συμβατότητα στα συστήματά μας. Το να λέμε ότι για μας αποτελείται χώρα πρότυπο σημαίνει ότι, ε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι είχατε ελεύθερες εκλογές. Αναγνωρίζουμε ότι οι εκλογές σας ήταν ελεύθερες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αναταραχές. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιασδήποτε εκλογικές αναμικρήσεις ανά τον κόσμο. Αλλά εάν εξετάσουμε όλες τις χώρες που έχουμε στην ανατολική μας συνεργασία, μπορούμε να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα είστε το υπαριθμόν ένα. Ε, και αυτό είναι σημαντικό, διότι ε, αναφερθήκατε στο δρόμο σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Μολδαβία. Ε, εγώ στο μέλλον βλέπω μάλλον δύο προσκόμματα και θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σα. Κατά πόσον καταρχά είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε τι μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τα επόμενα δυόμιση χρόνια, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτέ ε, μπορεί να είναι επώδυνε για του πολίτε, αλλά αν είναι επιτυχές, επιτυχής, ε, μπορούν και πάλι να είναι επώδυνε. Είστε διατεθειμένοι να το κάνετε αυτό διότι το δικαστικό σύστημα, το σύστημα των συντάξεων, τα θέματα αγοράς εργασίας ό,τι έχει σχέση με την εναρμόνιση ε, μεταξύ του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μολδαβικού συστήματος, διότι η επιλογή σας είναι να ε, έρθείτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως πρέπει να εναρμονίσετε τα συστήματά σας. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη δική μας την πείρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο δεν αναφέρατε κατά την άποψή μου και είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της υπερδυστερία. Υπήρχε πρόοδο προσφάτως και θα ήθελα να σας ρωτήσω ω υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, με αυτή σα την ιδιότητα και όχι με την ιδιότητα του αναπληρωτή Πρωθυπουργού, πώς βλέπετε το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Πέντε ή 2, σχέση σας με την Ουκρανία και τη Ρωσία για το θέμα αυτό. Πώς βλέπετε το όλο ζήτημα διότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε διατεθειμένοι να σας βοηθήσουμε. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένων Εθνών. Και γίνονται οι διαπραγματεύσεις στη Βιέννη, είμαστε παρατηρητές συνεχώς. Αλλά εσεί ε, πώ τη βλέπετε αυτή την προοπτική, κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, διότι εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσκομα για το μέλλον Έχουμε πει πείρα από το θέμα αυτό. Το να επιθυμεί κάποιο να είναι όσο το πιο κοντά γίνεται σε μια χώρα της Ευρώπης χωρίς να έχει επιλύσει πλήρως το θέμα των συνόρων του ε, με τους πιο κοντινούς του γείτονες. Και άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Δύσκολα τα ερωτήματα. Στη συνέχεια η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω ρουμανικά. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ στις Βρυξέλλες και επίσης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε τα όσα αναφέρει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο για την υπερνηστερία. Δεύτερη ερώτηση. Ε, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στην Ανατολική γειτονία και αν ε, προσφέρονται νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Next speaker. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Πρέντα, ε, από τη Ρουμανία και εκείνος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Συγχαίρω τη Μολδαβία για τις ε, πρόσφατες προόδους της. Τις αναφέρατε κι εσείς. Και κυρίως αναφερθήκατε στην τελευταία τριετία και κάνατε μια σύγκριση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς για τα γεγονότα και τις διαδηλώσεις του Απριλίου του 2009 στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Στο Κίσινο. Πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Έχουν υποστεί κυρώσεις εκείνοι ε, που βρέθησαν ένοχοι για την ε, βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη θλίψη της ε, και κατήγγειλε ε, αυτή την καταστολή εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών. Έχουν γίνει έρευνες, ήταν πάρα πολύ βαριές ε, οι κατηγορίες ή παραμένει ένα πέπλο μυστηρίου και θα πρέπει στο μέλλον να διαλευκανθεί. Στη συνέχεια, είδα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάνει πολύ αισιόδοξε προβλέψεις για το μέλλον της ε, μεγέθυνσης της οικονομίας. Πόθεν όμως θα προέλθει. Ε, από το 2013 ήδη και μετά περιμένετε βελτίωση, αλλά από πού θα έρθει αυτή στην οικονομία. Another click from Romania, Severin. Mr. Severin, please. Ο κ. Σεβερίν από τη Ρουμανία και πάλι. Ε, η υπερβολική δόση Ρουμαν... Ρουμάνων, ελπίζω όχι. Ε, θα μιλήσω στα αγγλικά για να με καταλάβουν και οι συνάδελφοι. Έχουμε ευκαιρίες να μιλάμε, μιλήσουμε στα ρουμανικά. Ε, με τον κύριο Λεανκά. Άκουσα τι ε, προτεραιότητε σα με πολύ προσοχή. Είναι σωστέ προτεραιότητε και θα πρέπει να υποστηριχτούν. Παρ' όλα αυτά, να προτείνω προσκέψη μερικέ άλλες ακόμα προτεραιότητε. Πρώτον, θα πρέπει να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο χώρο στην Μολδαβία έτσι ώστε να συμμετάσχει στην προσπάθεια όλη η κοινωνία και οι ηλικιωμένοι και όχι μόνο οι νέοι σε μια συζήτηση, ένα διάλογο για να καταλάβουν το project, ε, το, στόραμα όραμα της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμμετοχής της χώρας αυτήν. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ένας τέτοιος εσωτερικός διάλογος ε, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης θέματος των εθνικών ταυτοτήτων. Ε, δεύτερον, οι κοινωνικές προκλήσεις, τα κοινωνικά προβλήματα που δεν τα αναφέρατε. Ε, αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, όλες οι εξαιρετικέ ιδέες μεταρρυθμίσεων θα μπορεί να αποτύχουν. Και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ρόλο εδώ. Και τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να υλοποιήσετε μια στρατηγική ε, για να αντιμετωπίσετε τις ευρωπαϊκές προκαταλήψεις. Ίσως ήδη αναφερθήκατε σε ορισμένες από αυτές. Είπατε για παράδειγμα ότι η Μολδαβία είναι η πιο φτωχή χώρα της ε, Ευρώπης. Ε, ίσως με ορισμένους υπολογισμού, με βάση ορισμένους υπολογισμού να είναι έτσι. Αλλά πάντως ε, δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο ως η φτωχότερη ε, χώρα της Ευρώπης. Η Μολδαβία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει να προσφέρει στην Ευρώπη και στην οποία η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει πράγματα. Τελειώνοντας να σας ρωτήσω το εξή, να σα ζητήσω το εξή. Θα μπορούσατε να μα δώσετε λίγο περισσότερα ε, ε, σχόλια για τις απογοητεύσεις σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι αυτή, ποιε είναι αυτέ οι απογοητεύσει. Είστε ε, διπλωμάτης, οπότε ενδεχομένω θα μπορούσατε να ε, αναδιατυπώσετε με διαφορετικό τρόπο αυτή την ερώτηση, ίσως να μιλήσετε για, τις, ε, ε, για το τι αναμένετε εσείς, τις προσδοκίες σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, αντί να μιλήσετε για απογοητεύσεις. Mr. από την ομάδα των Πρασίνων. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ κι εγώ από πλευράς μου τον κύριο Λεάνκα ως προς τις πολιτικές εξελίξεις και τα όσα επέτυχε η κυβέρνησή σας και η χώρα σας. Όντως είναι μεγάλες οι πρόοδοι και εμείς τον αγνωρίζουμε. Σε ό,τι αφορά τον υποδειγματικό σας ε, ρόλο, είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες ε, προσδοκίες με την Ουκρανία και τη Γεωργία και απογοητευθήκαμε ικτρά. Ε, αυτή τη στιγμή το στατείτε εσείς στην ανάπτυξη και ελπίζω να είναι θετική αυτή εξέλιξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Δουβλίνο για την ε, υπερδνηστερία, αλλά χαίρομαι που επανήλθαν οι διαπραγματεύσει 5 συν 2 και έχει λίγο κατευναστεί το πνεύμα ως προ τα στρατιωτικά. Αλλά θέλει η Μολδαβία ε, ε, ή κάποιος άλλος εκεί στην περιοχή να δημιουργήσει ένα είδος ελεύθερη ζώνη στην υπερνηστερία, να γίνει ένα είδος Ταϊβάν και ε, φλερτάρει και η Ρωσία με την υπερδνηστερία για να δημιουργηθεί μια ευρασιατική οικονομική ένωση. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό. Τονίσατε επίση ότι ε, μεταφέρετε στην ομοθεσία σας ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές και ότι έχετε ακόμα δουλειά. Να σας αναφέρω το εξή τρία. Πρόσφατα περάσετε ένα νόμο κατά των διακρίσεων και δεν παίζει ρόλο καθόλου εκεί ο σεξουαλικός πολιτικός Μα και αυτό δεν θα πρέπει να είναι κριτήριο διακρίσεων, γιατί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρεται ε, αυτό, στη χώρα σας λείπει από την νομοθεσία. Επίσης μαθαίνω ότι σε έξι πόλεις και δύο περιφέρειες η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεστε περιορίζονται και καταπιέζονται. Εσείς πώς το αξιολογείτε και αυτό. Ευχαριστώ. Κολέγια Γκόμες, Κυρία Γκόμες, καλώς ήρθατε. Ε, σας συγχαίρω για, την πρόοδο. Για την πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα σας. Γνωρίζω τις ε, δυσκολίες. Ελπίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ότι είστε η πιο ε, φτωχή χώρα της Ευρώπης δεν θα πρέπει να σας εκφοβίζει. Αντιθέτως, εγώ προέρχομαι από την Πορτοκαλία, μια χώρα που παλιότερα θεωρείται και αυτή η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης και ενδεχομένως εξακολουθεί να είναι μία από τις φτωχότερες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει βελτιωθεί το βιωτικό μας επίπεδο κατά πάρα πολύ μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Ε, δεν αποτελεί αυτό κάτι που μας χωρίζει από τους υπόλοιπους. Το αντίθετο. Γνωρίζω επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και που συνδέονται με την υπερνηστερία και, την, και το, τη σύγκρουση εκεί γνωρίζω ότι βελτιώνει την κατάσταση. Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αναγνωρίζει κάποια πρόοδο στο δικαστικό σύστημα που επετεύχθη πέρσι. Οπότε είναι δυνατόν να προχωρήσετε αν ε, προσιλωθείτε σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα Αντί να σας ρωτήσω για τις, την απογοήτευση που νιώθετε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να το δω θετικά. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον πολιτικό τομέα, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε τα πολλά προβλήματα σχετικά με τα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαστικό σύστημα βέβαια εμπλέκεται, ελευθερία έκφρασης, ε, ανεκτικότητα, ε, ελευθερία έκφρασης, αλλά και ε, ανοχή ε, ομάδων όπως οι ομοφιλόφιλοι αλλά και άλλες ομάδες και με ανησυχεί επίσης η κατάσταση σε σχέση με το εμπόριο ανθρώπινης σάρκας. Ε, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για αυτό το, αυτά τα ζητήματα και τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Speaker, colleague ε, Ο κύριος Σιπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προφέρετε το όνομά μου. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να το πω. Θα μιλήσω πολωνικά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω. Να σας λέω Πρωθυπουργό, καλύτερο ακούγεται. Σας ευχαριστώ για την αποφασιστικότητά σας. για να υλοποιήσετε τις αλλαγές. Θυμάμαι όταν ε, ήταν οι εκλογές ε, του GCNOW, υπήρχε μια απεσιοδοξία εν γέννη. Ε, ήμουν παρόν ε, στις εκλογές και ξέρω πώς ήταν η διάθεση του κόσμου. Αλλά τελικώς από αυτή την απεσιοδοξία βγήκε αισιοδοξία και εσείς δείξατε αποφασιστικότητα. βεβαίως απομένουν πολλά πράγματα να κάνετε. Υπάρχει και αυτή η ψυχρή σύγκρουση με την υπερθυμιστερία Η ρήξη. Και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα ε, το λαό. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσετε όλες αυτές τις αλλαγές ε, ταυτόχρονα. Αλλά η ερώτησή μου αφορά κυρίως την υπερδυνιστερία. Ποιος θεωρείτε ότι είναι το ελάχιστο που θα μπορούσατε να αποδεχτείτε για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Αν δεν κάνω λάθος, η καλύτερη λύση για σας θα ήταν η υπερδυνιστερία να αποτελέσει ένα απόσπαστο τμήμα της Μολδαβίας. Αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερο ερώτημα. η δημόσια αποδοχή των μεταρρυθμίσεων. Το ακούσαμε και από άλλου. Εσείς σαφώς έχετε το στόχο την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε από την Πολωνία ότι ο λαός αυτό θα το υποστηρίξει υπό την προϋπόθεση ότι δεν τον επηρεάζει. Αυτή τη στιγμή όμως αυξάνεται η ανεργία, αυξάνονται οι τιμές ε, και ε, γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα των συντάξεων, ο κόσμος ανησυχεί. Με βάση την πείρα μας από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα αυτά που γνωρίζουμε για την Πολωνία. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει ώστε να μπορέσει ο κόσμος να υπερκεράσει τις δύσκολες αλλαγές. Ιδάλλον σας περιμένει ένας ε, δύσκολος δρόμος ε, ε, προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, κάποιος είπε ότι είχαμε μεγάλες προσδοκίες για κάποιες χώρες, αλλά ε, τελικώς ε, τα πράγματα έμειναν στάσιμα. Τι νομίζετε ότι μπορείτε να αντιλήσετε εσείς ως δίδαγμα από τις άλλες χώρες. Και θα ήθελα να συγχαρώ και τον ε, Μολδαβό διαμεσολαβητή στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος αποτελεί πρότυπο στην ανταλλαγή των πρακτικών ε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, μεταρρύθμιση των φωσοφρονιστικών καταστημάτων, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα με το διαμεσολαβητή της Πολωνίας και της Γαλλίας και αποτελεί ένα πολύ επιτυχές πρόγραμμα. Δεν αρκεί βέβαια να λέει κάποιο μόνο τι θέλει να επιτύχει. Καλό είναι να μαθαίνουμε και από όλου όσου έχουν περάσει ήδη τη διαδικασία. Και αν κάποιο την έχει περάσει, σα κατανοεί και καλύτερα. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ τους αδέλφους για τις πολλές και σημαντικές ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις. Και είμαι ικανοποιημένο γιατί βλέπω πως από τις ερωτήσεις πως κατανοείτε σε μεγάλο βαθμό πού βρισκόμαστε. Δείχνετε ενδιαφέρον για τη Μολδαβία και την όλη περιοχή και ε, οι ερωτήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι είσαστε πρόθυμοι και πρόθυμες να μας βοηθήσετε. Ας απαντήσω στις ερωτήσεις σας λοιπόν τώρα. Μόνικα, Μόνικα δεν έκανε ερωτήσεις, ε, μόνο σχόλια. Ο κ. Μπούζεκ έθεσε δύο ερωτήματα. Πόσο είμαστε έτοιμοι για τις μεταρρυθμίσεις, καταρχήν. Η αποφάση που πήρε το Κοινοβούλιο περασμένη Παρασκευή για τους δύο νόμους της αποφύγης των διακρίσεων και για την δημιουργία ενός πιο αυτόνομου οργάνου για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς ε, και θα ελέγχεται από το Κοινοβούλιο ε, κάτι που θα του δώσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτοί οι δύο νόμοι και μάλιστα ε, μέσω του δεύτερου νόμου ο διευθυντής ε, αυτού του οργάνου καταπολέμησης διαφθοράς ε, δεν θα διορίζεται, θα προκύπτει μετά από διαγωνισμό. Ε, αυτοί οι δύο νόμοι απέδειξαν την αποφασιστικότητα των αρχών της Μολδαβίας να προχωρήσουμε παρόλη την διαφωνία της αντιπολίτευσης και της ισχυρή προπαγάνδας. Έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια και πιστεύω ότι σε αυτά τα τρία χρόνια μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η Μολδαβία είναι μικρή χώρα και μερικές φορές το πιο μικρό είναι πιο όμορφο, αλλά όχι πάντα. Και μπορούμε να, να δείξουμε σε όλο τον κόσμο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ότι μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές και ε, θετικές σε ό,τι αφορά τη συντάξη του κόσμου, την ποιότητα ζωής, τους μισθούς και τις ελευθερίες. Περισσότερες ελευθερίες, για παράδειγμα ελευθερία μετακίνησης, ε, ελευθερία μετακίνησης χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δείξουμε ότι έχουμε ευρωπαϊκή προοπτική. Έχουμε πάρει την απόφαση αυτή και δεδομένου ότι έχουμε εξασφαλίσει τη σταθερότητα ε, δεν έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε το φάσμα νέων εκλογών, κάτι που σίγουρα θα δυσκόλευε ε, τις μεταρρυθμίσεις, οπότε μπορούμε να εστιάσουμε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες σας παρουσίασα. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μας ε, ικανοποιεί η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η δημοκρατία της Μολδαβίας ήδη από φέτος και για τα επόμενα δύο χρόνια παίρνει 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Είναι ένα πολύ, μια μεγάλη βοήθεια. Θα μας βοηθήσει γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα μας βοηθήσουν μόνο για τις μεταρρυθμίσεις αλλά και για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους και μας δημιουργούν και πίεση βέβαια. Δέχομαι και ζητώ από τους Ευρωπαίους ε, εταίρους μας ε, όχι μόνο να μας παρακολουθούν αλλά και να μας πιέζουν. Ευρωπαϊκή προοπτική σημαίνει ότι θα γίνουμε υποψήφοι, υποψήφια χώρα και η πίεση από τις Βρυξόλλες αλλά και από την κοινή μας νόμη, από την κοινωνία μας, θα μας δώσει περισσότερα κίνητρα σε κυβέρνηση και κοινοβούλιο να προχωρήσουμε. Είμαι σίγουρος για τον ενθουσιασμό μας και το ζήλο μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό. Δεν έχουμε και εναλλακτική λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να γίνουμε ευημερούσα χώρα. Σε άλλη περίπτωση θα χρειάζεται να συνεχίσουμε να ε, ε, μεταναστεύουμε σε άλλες χώρες, την Ιταλία, τη Ρωσία, τη Ρουμανία ή την Πορτογαλία για καλύτερη ζωή. Δεν έχουμε εναλλακτικέ λύσεις. Χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις και σε δύο χρόνια θα πρέπει να έχουμε αποδείξει στους πολίτες μας τη χρησιμότητα των μεταρρυθμίσεων αυτών. Για την υπερδυνιστερία ετέθησαν πολλές ερωτήσεις. κατά πόσον θέτει σε κίνδυνο την ενταξιακή μας προοπτική και τι πρόοδος έχει γίνει και ποιο είναι το μέλλον. ποιε είναι οι σχέσεις με την Ρωσία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ε, θα έχετε διαπιστώσει, αν παρακολουθείτε τι εξέλιξει, την θετική δυναμική. Ασφαλώς ακόμα απέχουμε πολύ από την ε, ε, οριστική λύση Είμαστε μακριά ακόμα και από το να πετύχουμε τις αρχές, να επισυμφωνήσουμε τις αρχές πάνω στις οποίες θα βασιστεί μια λύση. Όμως, χάρη στην θετική δυναμική, χάρη στην, ε, στο ζήλο της ε, νέας ε, κυβέρνησης είμαστε πολύ πιο κοντά πλέον. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα, μια αργή αλλά σταθερή επανενσωμάτωση αυτού του κομματιού της Μολδαβίας στην χώρα οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί. Καταφέραμε να ξαναξεκινήσουμε τις εργασίες των ομάδων εργασίας για τα τελωνία, την παιδεία, την καταπολέμηση του ρεωμένου εγκλήματος κλπ. Αυτό ε, δίνει αποτελέσματα, δίνει καρπούς. Κάποιος με ρώτησε ποιο είναι, ποιο, ποιο είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να δεχτούμε σε ό,τι αφορά την τελική λύση. Είμαστε ευέλικτοι. Είμαστε αρκετά ευελικτοί. Δεν λέμε ότι θα, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μια ομοσπονδία ή κάτι σύμφωνα με το βρετανικό μοντέλο ε, μια ε, ε, παροχή εξουσίας στην υπερνηστερία κλπ. Το κλειδί μιας οποιασδήποτε λύσης είναι η Μολδαβία να γίνει πιο ισχυρή ως κράτος δεν ε, θα πρέπει οποιαδήποτε λύση να μας βγάλει από, την, ε, από το δρόμο προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε λύση που ε, δεν θα αντιστοιχεί σε αυτό μας το όραμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή. Κανείς δεν θέλει μια δεύτερη Κύπρο, μια διχασμένη χώρα. και είμαστε σίγουροι ότι για να πετύχουμε το, το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, ε, ε, μάλλον το, η ύπαρξη αυτού του προβλήματος δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην χορήγηση του καθεστώτος υποψήφια χώρας. Γιατί λέμε ότι υπάρχει μια δυναμική, αλλά μόλις αποκτήσουμε και την προοπτική της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Γιατί ε, οι κάτοικοι τη υπερνηστερία θέλουν μια σταθερή, ισχυρή Μολδαβία. Ε, θέλουν να δουν την ζωή τους ε, πιο εύκολη μέσα στη Μολδαβία. Οπότε αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό σημείο, το σημείο κλειδί είναι να μας δοθεί αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική. Γιατί αυτό θα αποτελούσε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τη Μολδαβία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της και θα αποτελούσε ενθάρρυνση όχι μόνο για τους πολίτες της Μολδαβίας αλλά και σε, για ορισμένους από τους γειτονές μας. Ε, τώρα, για την σύνολο κορυφή του ΝΑΤΟ ασφαλώς ε, μας ικανοποίησε η αναφορά στην υπερνηστερία. Ε, ένα στοιχείο το οποίο δεν αναφέρθηκε μόνο, ε, μάλλον ε, ναι, είναι τα πυρομαχικά ε, τα οποία έχουν παραμείνει. Μια, αν είχε γίνει μια τέτοια αναφορά θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο. Ρωτήσατε επίσης για την ανατολική εταιρική σχέση. Ε, το Τσισινό επιλέχθηκε για την πρώτη συνάντηση των Υπουργών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα λάβει χώρα στις 5 Ιουνίου. Το διάλεξε η Κομισιόν. Ε, θα είναι και η κυρία Χέλγκερ Σμιτ και ο κύριος Φούλε. Και θα συζητήσουμε όχι μόνο διμερεί θέματα, αλλά και πολυμερή ζητήματα. Ε, έχουμε αργήσει, έχουμε μείνει πίσω. Ε, οι διαφορές στα πολιτικά συστήματα, οι φιλοδοξίε τη κάθε, το, κάθε χώρας μπορεί να είναι διαφορετικές αλλά ε, υπάρχουν και άλλα θέματα. Ε, πολιτική άμυνα, ε, πολιτική προστασία, συγγνώμη, φυσικές καταστροφές κλπ. που μπορούμε να συνεργαστούμε. από το 2009 και μετά, από τον Απρίλιο 2009 και μετά, δεν έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Πρέπει να, να, να προχωρήσουμε και ε, θα πρέπει το μυστήριο να πάψει ένα μυστήριο να διευκρινιστεί, να διαφωτιστεί ε, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, οι προβλέψεις είναι 3% μόνο. Για μας είναι χαμηλό ποσοστό. Ε, ελπίζω τουλάχιστον να πετύχουμε αυτό το στόχο του 3% μέσω ιδιωτικοποίησεων ε, ορισμένων ε, κρατικών πόρων θα μπορούσαμε ενδεχομένω να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κύριε Σεβερίν, κάνατε διάφορε ερωτήσει, προ, κοινωνικά προβλήματα. Έχετε δίκιο. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει, αλλά οι εκθέσεις αυτού του τύπου δείχνουν ότι η Μολδαβία πηγαίνει καλά. Είναι άξιοι άνθρωποι οι Μολδαβοί και αξίζουν καλή συμπεριφορά. Και η αρχή περισσότερα για περισσότερα θα πρέπει να μας φέρει εκεί που μας αξίζει. Οι προοπτικέ, ναι. Η βασική μας προοπτική είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Η βασική μας προσδοκία είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Έχουμε ε, το θέμα των θεωρήσεων, το θέμα της ε, εταιρικής σχέσης που έχει σχεδόν κλείσει. Για τις θεωρήσει ελπίζουμε ότι τις επομενε 9 9-10 μήνες θα έχουμε ε, λίστα τεχνικά προβλήματα ε, θα ήθελα να μας συμπεριφερθείτε όπως συμπεριφερθήκατε στην ε, Μακεδονία, Λεωμιλτή, Σερβία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Να μας δώσετε αυτό που αξίζουμε. Να μας επιτρέψετε, επιτρέψετε τους πολίτες μας να κυκλοφορούν ε, ελεύθερα χωρίς ε, πρόσθετους όρους. ήδη όροι που έχουν επιβληθεί είναι πιο αυστηροί από τους όρους που είχαν οι πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, ελπίζω θα τελειώσουν τα μέσα του επόμενου χρόνου και τις ε, διαπραγματεύσει για την ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών. Ελπίζω θα περάσουμε στις διαπραγματεύσει για την ένταξη. Ο κ. Σούλτς ε, ρώτησε για την Περνιστερία, αν θα μπορούσε να γίνει ειδική οικονομική ζώνη. ίσως έχουμε ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσει για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε μερικέ ζώνε ελεύθερων συναλλαγών στην ε, Μολδαβία. Και ε, στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προβλέπεται η λειτουργία τους για τα επόμενα 5-10 χρόνια μόνο. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δεχτεί ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα για την περνηστερία μονίμως. Αυτό που προσπαθούμε είναι οι, οι εκπρόσωποι τη της να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη συμμετείχαν στον πρώτο γύρο, θα έρθουν και εδώ στις Βρυξέλλες γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο να επωφελθούν από τη ζώνη ελεύθερων συνάργων με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, αυτοί εξαρτώνται από τις ευρωπαϊκές αγορές ε, περισσότερο από την η υπόλοιπη χώρα. Σε ό,τι αφορά την αποφυγή διακρίσεων και το αντίστοιχο νομοσχέδιο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ε, πετύχαμε ό,τι μπορούσαμε να πετύχουμε με δεδομένες συνθήκες. Ε, μην ξεχνάμε ότι... <laughs> Μην ξεχνάμε τι έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να, να φέρουμε την ε, νομοθεσία μας ε, να την ευθυγραμμίσουμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις, ευρω... τις ευρωπαϊκές οδηγίες δηλαδή. Στο άρθρο 7 του νόμου μας αναφέρεται, αναφέρονται ρητά τα δικαιώματα των ε, σεξουαλικών μειονοτήτων. Θα πρέπει τώρα να εστιάσουμε στην εφαρμογή αυτού του νόμου, να δημιουργήσουμε θεσμούς που θα μας οδηγούν σε μια ανεκτική και δημοκρατική κοινωνία. Ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρία Γκόμες μας ρώτησε για το θέμα αυτό. Αν δείτε την ε, έκθεση Freedom House που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Στην προηγούμενη περίοδο η Μολδαβία έκανε τεράστιο άλμα. Ε, μεγάλο άλμα ακόμα και αν συγκριθούμε με χώρες Δυτικών Βαλκανίων της Κεντρικής Ευρώπης. Και ασφαλώς έχουμε ακόμα σημαντικά πράγματα, για παράδειγμα την ε, ε καταπόλεμηση διαφθοράς Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Για την ελευθερία του τύπου, ε, ακόμα και εκεί κάναμε σημαντική πρόοδο. Από το 80 περάσαμε περίπου στο, στις 50. Θα, ε, βλέπετε το άλμα που έχουμε επιτύχει. Όμως θα συνεργαστούμε μαζί σας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε μια ένα θεσμοθετημένο διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητήσαμε. Τα 60, ένα κομμάτι των 60 εκατομμυρίων για το δικαστικό σύστημα θα αφιερωθεί όχι μόνο να αλλάξουμε την νοοτροπία των δικαστών, αλλά για να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λαθρεμπορίο ανθρώπων. Είμαι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για το θέμα αυτό πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα ε, είναι ντροπή. Είναι όνειδος. Έχει κοινωνικούς, ε, κοινωνικές και οικονομικές αιτίες. Ε, αν δείτε τα νούμερα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει σταθερή πρόοδος. Βέβαια έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και θα συνεργαστούμε με την κυρία Μάλστρομ και τον ειδικό εκπρόσωπό της σε την επόμενη εβδομάδα θα ε, έχουμε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του δικαστικού σώματος, ε, τους ε, κατατόπους εκπροσώπους του δικαστικού σώματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Έχουμε πρόοδο, θα συνεχίσουμε ελπίζω. Για την υπερνηστερία προσπάθησα να σας εξηγήσω ποιο είναι το ελάχιστο που μπορούμε να δεχτούμε. Για την... Ε, ε, βιάζομαι γιατί βλέπω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, γι' αυτό μιλάω γρήγορα. Πρέπει να δείξουμε στους ανθρώπους, στους πολίτες μας, ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ και ότι θα έχουν ωφέλη. Και ήδη έχουν κάποιο ωφέλη, αλλά σε δύο-τρία χρόνια πολύ μεγαλύτερα. Ε, ασφαλώς θα πρέπει να μιλήσουμε με την Πολωνία και τη Ρουμανία και άλλες χώρες για να διδαχθούμε από αυτές και να μικρύνουμε το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε. Όμως δεν ξεκινάμε τώρα. Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρέπει απλώς να ολοκληρωθούν. Ξεκινήσαμε με, την, με τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Χρειάστηκε να κλείσουμε σχολεία σε μικρά χωριά για παράδειγμα, αλλά με βοήθεια τη Παγκόσμια Τράπεζα, βάλαμε λεωφορεία και μεταφέρουμε του μαθητές στα, στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Χρειάζεται λοιπόν απτή βοήθεια και χρειάζεται και χρειάζονται και θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγγνώμη που καθυστέρησα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα τώρα. Thank you Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Εξαιρετική. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσά και στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ στο επανειδή.